Thank you very much for being patient with me. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήρθανε. Μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά έχουμε μεικτή συνεδρίαση δύο επιτροπών. Με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν. Ως ε, τρίτη αντιπρόεδρος μου ζητήθηκε να προεδρεύσω και χαίρομαι γιατί έχουμε μία σημαντική σήμερα επέτειο. Έχουμε δύο χρόνια από την κοινή πορεία για το μέλλον που είχαμε συνυπογράψει τότε περιμένοντας τον κύριο Αουστριβίτσιους, τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τις συστάσεις και με την εισαγωγή μου. έγινε μια πρώτη κοινή συνεδρίαση πέρσι και συνεχίζουμε ακριβώς λόγω αυτής της ε, κοινή πορείας όπως λέγεται επιπλέον έχουμε συχνά συνεδριάσεις λόγω της ε, νομοθετικής μας αρμοδιότητας για το θέμα των παρανόμως διαμενών των υπηκών τρίτων χωρών και η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών μας ενημέρωσε για όλες τις ε, συμφωνίες επανεισδοχής ε, καθώς ακριβώς εξετάζουμε το θέμα του κοινού, της κοινής πορείας με το Αφγανιστάν. Οι συμφωνίες επανεισδοχής βασίζονται στο άρθρο 230 και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα συνένεσης. Και αυτό βεβαίως περιλαμβάνει και δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου και εξέτασης της εφαρμογής τους για την Επιτροπή Λίμπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διαρθρωμένη παρακολούθηση όλων των συμφωνιών, επισήμων ή ανεπισήμων. Η κοινή πορεία για το μέλλον με το Αφγανιστάν ήταν η πρώτη τέτοια ανεπίσημη ή όπως τους λέει η Κομισιόν διευθετήσεις. Και μετά την κοινή πορεία για το μέλλον ακολούθησαν και άλλες τέτοιες συμφωνίες με την Αιθιοπία, τον Μαγκλαντές, την Γουινέα και την Γκάμπια. Οι εξελίξεις αυτών των διευθυντήσεων είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαιτέρως ε, την Επιτροπή μας καθώς μπορεί έτσι να στερηθεί το Κοινοβούλιο της αρμοδιότητας του άρθρου 218 συγκεκριμένα. Η Επιτροπή μας θεωρεί ότι πέραν από τις επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής οποιοδήποτε άλλο τέτοιο έγγραφο ή δήλωση για τις επανεισδοχές πρέπει να εξετάζεται. Ιδιαιτέρως όταν παράγει αποτελέσματα ε, ισοδύναμα ή παρόμοια με τις συμφωνίες αυτές για τον σκοπό αυτό. Η πρόσβαση στο κείμενο της συμφωνίας έχει μεγάλη σημασία η Κομισιόν μας είπε ότι το κείμενο της συμφωνίας με την Αιθιοπία, Γουινέα και την ε, Γάμπια δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί αυτήν τη στιγμή ανταυτού. Η Κομισιόν προτείνει να υπάρξει μια συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών που θα μας δείξει το κείμενο των συμφωνιών τις οποίες έχει συνάψει δηλαδή με τον Μπαγκλαντές, Αιθιοπίας και Γαμπής. Αυτό της Αιθιοπίας έχει διαρρεύσει, το διάβασα και ε, είναι το ίδιο με την κοινή πορεία για το μέλλον. Δηλαδή ένα από τα πρώτα άρθρα λέει δεν είναι νομικό κείμενο το παρόν, οπότε δεν προκύπτουν από αυτό δικαιώματα. Είναι αδιανόητο, δηλαδή να υπάρχει μια συμφωνία εντός του Συμβουλίου με τα κράτη-μέλη και να μην το λέμε συμφωνία και να μην είναι νομικό κείμενο. Και για να γίνω πιο σαφής, είναι απολύτως απαραίτητο να γίνουν σεβαστές οι υποπτικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρα οι εξελίξεις αυτές δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περιορίσουν το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και για όλους αυτούς τους ε, λόγους ε, θεωρώ πως η κοινή πορεία για το μέλλον με το Αφγανιστάν έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι η πρώτη σημασία του Ιουδιστού και δυστυχώ το μόνο κείμενο ανεπίσημης συμφωνίας στο οποίο το Κοινοβούλιο είχε επίσημη πρόσβαση. Οπότε θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε σήμερα μια λεπτομερή ενημέρωση για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και το πώς η συνεργασία αυτή έχει εξελιχθεί στην πράξη στο πλαίσιο της γενικότερης μεταναστευτικής πολιτικής ε, της Ένωσης. Επ' αυτού, λοιπόν, και χαίρομαι που έχει έρθει ο κύριος Αστρεβίτσιος, επικεφαλής αντιπροσωπής με το και του δίνω το λόγο. Συνάλφοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που διεξάγεται αυτή η κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνη και Ασφάλειας. Χαίρομαι για αυτή τη συνεργασία με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Είμαι πεπισμένο ότι οι επιτροπές και οι αντιπροσωπείες αλληλοσυμπληρώνονται και μπορούν να συνεργάζονται. Δεύτερον, χαίρομαι που μας δίνεται ξανά η ευκαιρία να συζητήσουμε μετά, τον μετά την τελευταία μας φορά το Δεκέμβρη του περασμένου έτους το θέμα του Αφγανιστάν. Ελπίζω ότι θα το επαναλάβουμε και στο μέλλον. Πριν δώσω το λόγο στους ε, καλεσμένους μας, θα ήθελα να κάνω κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις. Φαίνεται λογικό να δούμε τα σημερινά νούμερα για να καταλάβουμε ποιε μπορεί να είναι οι απειλέ και ποιο είναι το πρόβλημα. Σύμφωνα με τα στατιστικά τη ΥΠΑ τη Αρμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε, 12.052 Αφγανοί πρόσφυγε επέστρεψαν στο Αφγανιστάν φέτο μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι 75% λιγότερο ε, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 48.055 πρόσφυγες είχαν επιστρέψει στο Αφγανιστάν την ίδια περίοδο πέρσι. Από τους 12.052 που επέστρεψαν φέτος στο Αφγανιστάν, 10.275 ε, ε, ήρθαν από το Πακιστάν. 1966 ε, από το Ιράν και μόνο 111 από τρίτες χώρες. Από το 2002, όταν πάνω από 1.800.000 πρόσφυγες επέστρεψαν στο Αφγανιστάν, ο αριθμός των επιστρεφόντων μειώνεται συνεχώς. Εκτός από το 2016, όπου 370.000 επέστρεψαν στο Αφγανιστάν. Αυτά τα νούμερα καταδεικνύουν την κατάσταση της ασφάλειας στη χώρα αλλά και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, παράδειγμα στέγαση, απασχόληση κλπ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε την κατάσταση στη χώρα πριν αποφασίσουμε το πώς και το πότε στέλνουμε ανθρώπους πίσω. Τώρα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον πρώτο μας ομιλητή, ο κ. Ιωάνν Ντράγκος Τοντορέτσι. Είναι ε, ε, της, ε, ε, του τμήματος παράτυπης μετανάστευσης. Θα σας δώσω 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω αναφερόμενος στο θεσμικό ζήτημα το οποίο ετέθη στην αρχή. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν πολλές φορές. Έχουν ανταλλαγεί επιστολές ανάμεσα στον πρόεδρο της ΛΥΜΠΕ και την ε, Κομισιόν, για παράδειγμα. Πρέπει να το δούμε και από νομικής και από πολιτικής και θεσμικής πλευράς. Εμείς έχουμε επαναλάβει τη θέση μας πολλές φορές και ποια είναι αυτή η θέση και από, ότι και από νομικής πλευράς η θέση μας είναι πως Αυτές δεν είναι συμφωνίες που έχουν νομική ισχύ, γι' αυτό το λόγο το άρθρο 18 δεν εφαρμόζεται. Αντιλαμβανόμαστε ότι το Κοινοβούλιο θέλει να λαμβάνει εκθέσεις, ε, επιζητεί τη διαφάνεια και επιθυμεί να ελέγχει το περιεχόμενο και την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. για αυτό το λόγο ερχόμαστε τακτικά στην Επιτροπή ή στέλνουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας σε ό,τι αφορά το στάδιο των διαπραγματεύσεων και όποιες διευθετήσεις ε, γίνονται για την εφαρμογή. Η, η πρόεδρος αναφέρθηκε στη τελευταία συνάντηση στο τέλος Ιουνίου. Μετά από αυτήν σας ενημερώσαμε. Κατόπιν επιστολής του Πρόεδρου Μωράης στον Επίτροπο Αβραμόπουλο, εστάλει πριν από μία εβδομάδα νομίζω επίσημη απάντηση όπου προτείναμε ένα πολύ συγκεκριμένο μηχανισμό επί τη βάση του οποίου θα μπορούσαμε να θέτουμε στην διάθεση των ενδιαφερόμενων μελών πληροφορίες σύμφωνα με το μηχανισμό των εκθέσεων σεβάλ. Αυτοί δηλαδή, αυτά τα μέλη τα οποία επιθυμούν να λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση, θα μπορούν να το κάνουν και να τη συζητούν μαζί μας. Αυτό είναι το θεσμικό. Τώρα, για την συνεργασία με το Αφγανιστάν για θέματα μετανάστευσης και για ζητήματα επιστροφών. Πάντοτε λέγαμε ότι ο διάλογος για το μεταναστευτικό με το Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Βασίζεται σε δύο βασικές αρχές. Πρώτον, η περιφερειακή προσέγγιση και δεύτερον, η σφαιρική προσέγγιση. Περιφερειακή προσέγγιση διότι αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Αφγανιστάν μέσα στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Υφίσταται ανάγκη να αντιμετωπιστούν και οι εσωτερικοί εκτοπισμοί και όλες οι μετακινήσεις ε, στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει το Αφγανιστάν. Δεύτερον, σφαιρική προσέγγιση. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο για το Αφγανιστάν. Έχουμε προσπαθήσει σε, να το ενσταλάξουμε στους διαλόγους με όλες τις χώρες με τις οποίες συζητάμε. Θέλουμε να δούμε όλες τις πτυχές της μετανάστευσης και να οικοδομήσουμε ένα διάλογο, ένα μηχανισμό συνδρομής με την κάθε χώρα, με τους εταίρους μας σε αυτή την ε, χώρα, για όλες αυτές τις πτυχές της μετανάστευσης. Τώρα, για, το, ε, για την κοινή πορεία για το μέλλον. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Αφγανιστάν. Ε, τυπικά Και πάλι δεν πρόκειται για νομική συμφωνία. Πρόκειται για μια δέσμευση. Πολιτική δέσμευση. Και δεν απορρέουν από την κοινή πορεία για το μέλλον ε, κάποιες καινούριες υποχρεώσεις. Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι επιστροφές μπορούν να γίνουν με προβλέψιμο και διαρθρωμένο τρόπο. Προβλέψιμο με την έννοια του ότι θα το γνωρίζουν οι ίδιοι, οι επιστρεφόμενοι και οι αρχές από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αφγάν, Αφγανιστάν και Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα τελευταία λεπτά των, της ομιλίας μου να σας πω για τα μέτρα επανένταξης τα οποία έχουν ληφθεί και τα οποία ακολουθούν και συνοδεύουν τις επιστροφές. όλες, για, σε όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες επανειστοχής ε, είναι απόλυτο απαραίτητη επανένταξη έτσι ώστε η διαόλια διαδικασία να είναι βιώσιμη. Σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν δε έχουμε κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ασφαλείας στο Αφγανιστάν. Δεν είναι η πιο εύκολη περίπτωση. Αυτό το αναγνωρίζουν και οι ίδιες οι αρχές που αποφασίζουν την επιστροφή και την διατάσσουν. Εξετάζοντας τις προσπάθειες επανένταξης, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ένα πολύ καλό project που αντιμετωπίζει πολλές διαστάσεις της επανένταξης. Καταρχήν έχουμε την κοινωνική διάσταση τη διάσταση της τοπικής κοινωνίας. Μην ξεχνάμε στο Αφγανιστάν υπάρχουν ε, αστικές και εξωαστικές περιοχές. Για τις δεύτερες ε, προβλέπουμε συστήματα άδρευσης για τις περιοχές αυτές, θερμοκήπια τα οποία εγκαθιστούμε ήδη τώρα και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι επιστρέφοντες τα επόμενα, τους μήνες για αυτές τις αγροτικές περιοχές ε, έχουμε 1962 ε, επιστρέφοντες και 1200 οικογένειες που τους φιλοξενούν. Προβλέπουμε επίσης ε, προσωπική βοήθεια και σε αστικές περιοχές, σε πόλεις, ε, με δάνεια, ε, εγγυήσει ε, κλπ. Η Ράντα είναι η υπηρεσία η οποία είναι ο πάροχος αυτής της βοήθειας Ε, και οι διαδικασίες προσαρμόζονται στις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας. Στις πόλεις ε, θέλουμε να στηρίξουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου πραγματικά να βοηθήσουμε την βιωσιμότητα της επανέντεξης. Επίσης κατάρτιση και τεχνική συνδρομή σε επιστρέφοντες. Έχουμε εντοπίσει 73 κέντρα εκπαίδευσης με επιμόρφωσης τα οποία χρησιμοποιούνται στις, ε, ε, στην υλοποίηση των σχεδίων μας. Επίσης, στείλουμε και κέντρα ενημέρωση για την επανένταξη. Εξετάζουμε την Κουντάρ, τη Λάγμαν και την Καμπούλ ως περιοχές προτεραιότητας. Αυτά είναι όσα έχουμε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια ελπίζω να καταλαβαίνετε τη σημασία την οποία δίνουμε στην επανένταξη. Ευχαριστώ. Thank um, Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σαμίρα Χαμίδη από την ε, Διεθνή Αμνηστία που σας συνάντησα νωρίτερα σήμερα που έχει ένα εξαιρετικό βιογραφικό. Έχει εργαστεί και εντό του Αφγανιστάν για τα δικαιώματα των γυναικών και τώρα είναι υπεύθυνη για την περιφερειακή εργασία της αμνηστίας εντός και γύρω από το Αφγανιστάν. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά παρακαλώ όχι πάνω από 10 λεπτά γιατί θέλω να έχουμε χρόνο για ερωτήσεις και θα πω ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα ήθελα στην συνέχεια όταν θα απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας υποβληθούν να είστε πολύ συγκεκριμένος είτε θα μιλάτε για ενσωμάτωση ε, ε, ανθρώπων που έρχονται από την Ευρώπη και άλλους που έρχονται από αλλού, ποιο διευθύνει τα προγράμματα και τι προπολογισμοί χρησιμοποιούνται για αυτά όλα γιατί είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Κυρία Χαμίντη, έχετε το λόγο. πρέπει να πιέσετε το κομβίον. Για να ανάψει το μικρόφωνο σας. Ναι. Πρέπει να σας ακούμε για να σας μεταφράζουν οι διερμηνήσεις. Καλησπέρα σας και πάλι και ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να σας απευθύνω σήμερα το λόγο. Να σας ευχαριστήσω την ΕΕ Επιτροπή που καλέσατε τη Διεθνή Αμνηστία και μας δίνει την ευκαιρία να σας μιλήσουμε για όλα τα προβλήματα που που αντιμετωπίζουμε και κυρίως για την κοινή πορεία για το μέλλον. Κυρίες και κύριοι, στο Αφγανιστάν ε, πρόκειται για μια κρίσιμη φάση. Η ευκαιρία που εμφανίστηκε από το 2001 για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την δίκαιη ανάπτυξη, τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, καθώς και για τη συμμετοχή των νέων και των γυναικών ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Οι Αφγανοί είναι προσιλωμένοι στο να εργαστούν για θετικές εξελίξεις στην χώρα και συμβάλλουν γιατί αναζητούν ε, την παιδεία, ε, ε, συμμετέχουν σε εκλογές, συμμετέχουν σε δίκτυα υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ωστόσο, δεν είναι πολύ εύκολη η πραγματικότητα. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε μετά από 17 χρόνια στήριξη. Η αλήθεια είναι πως καθημερινά επιδεινώνεται η κατάσταση στη χώρα. Η κατάσταση της ασφάλειας έχει επιδεινώσει επιδεινωθεί. Δεν μπορεί να δεχτεί κανείς επίθεση σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Η... Τα αντικυβερνητικά στοιχεία επιτίθενται εναντίον σχολείων, εγκαστιατορίων, νοσοκομείων, ε, τζαμιών ακόμα και ε, εναντίον ε, γκαλερί τέχνης. Βρίσκουμε πως μηνιαία γίνονται τουλάχιστον δύο ε, τρομοκρατικές επιθέσεις και έχουμε φτάσει σε νέο ρεκόρ όσον αφορά τα θύματα 1.692 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέχρι τον Ιούλιο ε, του τρέχοντος έτους. Ε, μόνο τους πρώτους έξι μήνες δηλαδή του τρέχοντος έτους. Να σας δώσω παραδείγματα. Πριν από δύο μήνες ένα ε, πανεπιστήμιο δέχτηκε επίθεση όπου 24 φοιτητές από τα 16 μέχρι τα 20 σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν. Ένας, ένα, μια αθλητική οργάνωση δέχτηκε επίθεση και ένας 28χρονος δημοσιογράφος που μιλούσε πέντε γλώσσες και είχε μεγάλες ελπίδες στην περιοχή ε, σκοτώθηκε στη διάρκεια αυτής της επίθεσης. Δυστυχώς η αφγανική κυβέρνηση δεν καταφέρνει να προστατεύσει τους πολίτες της. Επίσης δεν μπόρεσε να στηρίξει ούτε τα θύματα αυτού του πολέμου που σοβεί στο Αφγανιστάν. Οι περισσότεροι Αφγανοί αντιμετωπίζουν τεράστια φτώχεια λόγω έλλειψη στήριξη. Είναι επίση εκτοπισμένοι στην ίδια του τη χώρα. 1,1 εκατομμύριο είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι σε ολόκληρη τη χώρα λόγω συνεχιζόμενων συγκρούσεων. Είναι σημαντικό λοιπόν να θέσουμε το ερώτημα πόσοι από πιστεύετε πραγματικά και ανησυχείτε πραγματικά για την ασφάλεια όσων θέλουν, ότι θέλετε να, να επιστρέψετε στο Αφγανιστάν. Ακόμα και μέσω αυτού του υποτιθέμενου μηχανισμού επιστροφών όπου υποτίθεται ότι γίνονται θελοντικές επιστροφές. Διάβασα για τα ζητήματα το, τα όσα λέγονται για το Αφγανιστάν ε, ε, δεν αναφέρεται όμως εκεί καθόλου η ασφάλεια και η προστασία των ε, Αφγανών κρατούμενων. Στην ουσία όταν επιστρέφετε ανθρώπους στο Αφγανιστάν τους στέλνετε πίσω στον κίνδυνο. Θέλω να θυμίσω τις συστάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας όσον αφορά την επιστροφή Αφγανών από την Ευρώπη επί τη βάση μιας ε, έρευνας που εμείς ξεκινήσαμε το, και κάναμε ε, από τον Οκτώβριο του περασμένου ε, έτους. Αν και η κοινή πορεία για το μέλλον ε, μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν είναι υπό, εξε, εξέλιξη, θα πρέπει να είναι, ε, έχετε υπόψη ότι κανένα Αφγανό δεν πρέπει να σταλεί εκεί μόνο και μόνο επειδή η μεταναστευτική πολιτική τη Ευρώπη είναι να αυξηθούν οι επιστροφέ με οποιοδήποτε κόστο. Αυτό. Αυτό το επιχείρημα πρέπει να αμφισβητηθεί. Δεν αντιμετωπίζει την ασφάλεια των Αυγανών. Ε, επίσης είναι, πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή η συμφωνία. Η Διεθνής Αμνηστία κάνει έκκληση για την αναστολή των επιστροφών των Αυγανών μέχρι, ότου να επιτρέψει η κατάσταση στη χώρα την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή αυτών των ανθρώπων. Η παρακολούθηση διαρκής για, επίσης για την κατάσταση των επιστρεφόντων με, και πρέπει να συμπεριληφθεί στη νέα κοινή πορεία για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήρης έλλειψη πρόσβασης στις πληροφορίες για το τι συμβαίνει σε όσους επιστρέφονται στο Αφγανιστάν. Παρακαλώ, να θυμάστε ότι πουθενά δεν υπάρχει ασφάλεια. Είναι άδικο να αποφασίζετε ε, ε καθήμενοι εδώ να στείλετε κόσμο ακόμα και στο νότιο Αφγανιστάν η είπατε αρμοστία για τους πρόσφυγες και οι, οι, οι, οι γραμμές για την προστασία των προσφύγων πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως. Η Καμπούλ δεν είναι ε, ε, ασφαλής, μέρο, ασφαλές μέρος για να επιστρέφονται οι πρόσφυγες. Πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση επιτόπου με βάση τις ενημερώσεις από τους ανθρώπους που βρίσκονται και εργάζονται επιτόπου ολόκληρο το χρόνο. Εγώ θα ήθελα να κλείσω ε, τονίζοντας ότι οι Ευγανοί δεν αξίζουν αυτό που αντιμετωπίζουν σήμερα. Όπως και εσείς θέλετε να ζείτε με ασφάλεια μαζί με τις οικογένειές σας, αφήστε και εκείνους να το καταφέρουν αυτό. Μην τους αναγκάζετε να επιστρέψουν στο Αφγανιστάν στον κίνδυνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε ερωτήσεις. Ε, βλέπω την κυρία Σπινέλη. και μετά τον κύριο Αουστρεβίτσιους. Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ. Άκουσα την παρέμβαση της Επιτροπής που περιέγραψε το κοινή πορεία για το μέλλον ως μια ατζέντα για επιστροφές, παναπατρισμούς που βασίζεται σε διαρθωτικές και προληπτικές ε, πολιτικές. Άκουσα την περιγραφή σας για τις ε, πρωτοβουλίες επανένταξης των ε, Αφγανών στην χώρα τους και δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι ικανοποιητική καμία από αυτές τις περιγραφές και αυτές τις διαβεβαιώσεις εφόσον ε, στην πράξη βλέπουμε να επικρατούν άλλα ε, σε συνθήκες αυτό που περιγράφει δηλαδή η Διεθνής Αμνηστία αλλά και που το γνωρίζουμε όλοι μας και η Κομισιόν το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Η πραγματικότητα σε σχέση με τους επαναπατρισμούς και την ένταξη αυτά λένε το 72% Δηλαδή τα δύο τρίτα των Αυγανών που επαναπατρίζονται επιλέγουν αμέσως μέσα σε λίγες εβδομάδες ε, επιλέγουν αμέσως πάλι το δρόμο της φυγής. Δεύτερη πραγματικότητα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μετά από την κοινή πορεία για το μέλλον ε, πολλαπλασιάστηκαν οι επαναπατρισμοί επί τρία τα τελευταία τρία χρόνια πρώτη είναι η Νορβηγία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία. Και οι απελάσεις γίνονται πλέον μαζικά. Στη Γερμανία 68 οι απελάσεις, μεταξύ των οποίων ένας νέος 23 ετών που αυτοκτόνησε. Ναι, μια στιγμούλα μόνο παρακαλώ, γιατί σπάνια μιλάμε για το Αφγανιστάν. Εμείς, οι πολλές χώρες, σε βάση περιπτώσει μέλη, ε, συμμετέχουν σε, μια, σε έναν αποτυχημένο πόλεμο από το 2001, χρόνια και χρόνια δηλαδή, και δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουμε να κοιτιόμαστε στον καθρέφτη χωρίς να τρεπόμαστε υιοθετώντα ε, τέτοια πολιτική επαναπατρισμού όπως αυτή που περιγράφεται στην κοινή πορεία για το μέλλον. Λυπούμε που μιλάω με σκληρά λόγια, αλλά θα ήθελα να έχω απαντήσεις. Thank ευχαριστώ, Μπάρμπαρα. Ε, συμφωνώ, αλλά ε, η Προεδρία οφείλει βεβαίω να ακούσουμε και απαντήσεις πριν έρθει ο κύριος Αβραμόπουλος. Λοιπόν, Αυστρεβίτσιους και για Ένα λεπτό. Εντάξει, Τσούντιθ. Λοιπόν. Η ερώτησή μου προς τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για τα άτομα τα οποία έρχονται από το Αφγανιστάν υπάρχει κάποιο σχέδιο να αλλάξει η στήριξη που τους δίνουμε σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμη η εμπειρία που έχουμε και αν θα συνεχίσουμε. Και το ερώτημά μου προς την κυρία Χαμίντη είναι το εξής. Όσοι επιστρέφουν, ε, κάτι έχουν μάθει και το διαδίδουν. Πώς θα περιγράφατε την γενική διάθεση και σε ποιο βαθμό αυτό προκαλεί σε άλλους να επιστρέψουν μόλις μάθουν ε, το τι συνέβη στους προηγούμενους. Κύριε Φόχητ, να ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι στην Ευρώπη έχουμε 100.000 άτομα που ε, έχουν ζητήσει άσυλο και έρχονται ε, υπό διάφορα προσχήματα. Αλλά στο Αφγανιστάν, εκεί πέρα, το ΝΑΤΟ κάνει την δουλειά του, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων. Οπότε εγώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ακριβώς εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πιεζόμαστε ε, να επιστραφούν οι Αυγανοί, δηλαδή ακόμα και οι παλιοί απικιοκράτες όταν έφευγαν από μια χώρα έπαιρναν κάποια άτομα μαζί τους ή προσπαθούσαν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους. Έχουμε συνεργαστεί δηλαδή με κάποια άτομα και ακριβώς ε, ούτε αυτά τα άτομα δεν ε, φέρνουμε πίσω. Αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα είμαι σύντομη, γιατί ένα από τα πρώτα ερωτήματα τα οποία είχαμε θέσει είναι γιατί έχουμε κοινή πορεία για το μέλλον με το Αφγανιστάν. Κάτι το οποίο ξεκίνησε σε μια στιγμή που αυξανόταν η βία και η κατάσταση γινόταν χειρότερη. Γιατί λοιπόν έχουμε κοινή πορεία με το Αφγανιστάν και όχι κοινή πορεία με το Μαρόκο, ξέρω εγώ. Αυτή είναι μια ερώτηση. Ισχύει ότι ίσως ήταν δυνατόν να ασκηθεί πίεση στο Αφγανιστάν για να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει το ίδιο με άλλες χώρες για να συμφωνήσουν κάτι τέτοιο. Δεύτερη ερώτηση. Τι ξέχασα τώρα. Οπότε θα σταματήσω εδώ. Ο κύριος Ντόρφμαν. Να ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα βεβαίως την συνάδελφο Πινελή. Δεν ξέρω αν έχει πάει στο Αφγανιστάν και στην Καμπούλ συχνά, μάλλον όχι πολύ συχνά. Εγώ είχα πάει όμως στο τελευταίο ταξίδι της αντιπροσωπείας με τον κύριο Αουστρεβίτσιους. Μια ολόκληρη εβδομάδα περάσαμε στην Καμπούλ και το ε, κοινωνικό πρόβλημα στην Καμπούλ δεν είναι οι επιστροφές από την Ευρώπη. Αυτό μας το είπε και ο Πρωθυπουργό. Είναι ε, δευτερεύον εντελώς. Δεν απασχολεί την κυβέρνηση. Το πραγματικό πρόβλημα στην Καμπούλ και στο Αφγανιστάν είναι οι μαζικές επιστροφές από το Πακιστάν όπου εκατοντάδες χιλιάδες άτομα διώκονται από το Πακιστάν, επιστρέφουν στο Αφγανιστάν και αυτό δημιουργεί εκρηκτική κοινωνική κατάσταση και τους βλέπει κανείς σε ολόκληρη την πρωτεύουσα. Και μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος κρατάει εδώ και 50 χρόνια σχεδόν. Οπότε η ερώτησή μου είναι υπάρχουν κάποιες επαφές της ε, Κομισιόν ή άλλων με την πακιστανική κυβέρνηση γιατί νομίζω ότι αυτό το οποίο θα βοηθούσε όντως το Αφγανιστάν είναι να σταματήσουν αυτές οι μαζικές επιστροφές ε, από το Πακιστάν. Και έτσι ακριβώς ε, να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν με κανέναν τρόπο στην ε, Καμπούλ ε, να μην ε, βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Έβαλα και εμένα τον κατάλογο και έτσι τελειώνουμε και μετά θα ακούσουμε την Κομισιόν. Και την κυρία Χαμίντη. Βρήκα εδώ πέρα την αρχική κοινή πορεία για το μέλλον πριν από δύο χρόνια και θα ήθελα να καταλάβω κάποια πράγματα. Η κοινή πορεία για το μέλλον ξεκαθαρίζει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν θα επιστρέφονται χωρίς να έχουν εντοπιστεί τα μέλη της οικογένειάς τους ή κάποιες διευθετήσεις για να τους υποδεχτούν στο Αφγανιστάν. Από την κοινή πορεία διαβάζω. Η κοινωνία των πολιτών ε, όμως μας λέει άλλα. Ότι δεν βρίσκουν τις οικογένειες και ότι ε, δεν υπάρχει επανένταξη. Και μάλιστα η προστασία των ανηλίκων υπάρχει στα χαρτιά στο Αφγανιστάν αλλά δεν λειτουργεί. Πώς μπορεί η Κομισιόν να εγγυηθεί ότι θα σεβόμαστε αυτό το άρθρο τη κοινή πορεία για το Το άλλο λέει τα προγράμματα επιστροφή και η βοήθεια επανένταξη είναι κάτι το ξεχωριστό από την βοήθεια την αναπτυξιακή που παρέχεται στο Αφγανιστάν. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ε, στις εξηγήσεις που δώσατε πριν ε, ποια από τα έργα τα οποία αναφέρονται είναι εκτός του αναπτυξιακού προπολογισμού και ποια είναι του αναπτυξιακού προπολογισμού. Και αν δεν μπορείτε τώρα να μου το πείτε μετά γραπτός. Επίσης η κοινή πορεία για το μέλλον αναφέρει την δυνατότητα να φτιαχτεί ένα ξεχωριστό τερματικό κτίριο στο αεροδρόμιο της Καμπούλ για τις επιστροφές έχει γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Και όλα αυτά τα ρωτάω γιατί προσπαθούμε ακριβώς να ελέγξουμε την κατάσταση και το θέμα εδώ πέρα της κοινή πορείας για το μέλλον. Δεν είναι τόσο πολύ το κομμάτι της αναπτυξιακής βοηθείας που αφορά η Επιτροπή, αλλά το κομμάτι των επιστροφών, ε, για το οποίο είναι πολύ λεπτομερής η κοινή πορεία για το μέλλον. Λοιπόν, το λόγο έχει με μετά κυρία Χαμίντη. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εντάχει σε όλες τις ερωτήσεις. Πρώτον, γιατί κοινή πορεία για το μέλλον με το Αφγανιστάν. Γιατί τα κράτη-μέλη είχαν ε, συμφωνήσει συνενετικά ότι κάτι έπρεπε να γίνει με το Αφγανιστάν, ότι χρειαζόταν μια συμφωνία. Και εμεί ακολουθήσαμε αυτή την πολιτική δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη-μέλη και ε, ξεκινήσαμε διαπραγματεύσει. Πώ μπορούν να γίνουν επιστροφέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ το Αφγανιστάν. Θα επαναλαμβώ αυτό που είπα προηγουμένως αλλά και παλιότερα. Καμία επιστροφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται χωρίς να έχει γίνει σύμφωνα με τον νόμο η ε, απαραίτητη ατομική εξέταση. Εξετάζουμε όλες τις πτυχές κάθε υπόθεση χωριστά. Κοιτάξτε τα νούμερα. Τα νούμερα είναι εύγλωτα σε ό,τι αφορά τις επιστροφές από την Ευρώπη. Είναι πολύ λιγότερες από ό,τι αναμέναμε ή φοβόμασταν το 2016. Από τότε η Frontex έχει κάνει 700 καταναγκαστικές επιστροφές. Οι περισσότεροι επιστρέφοντες προέρχονται από τις γειτονικέ χώρες και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση η στήριξη που δίνουμε δεν το λαμβάνει υπόψη αυτό. Γιατί από την αρχή θελήσαμε να βοηθήσουμε το Αφγανιστάν στην προσπάθεια που κάνει η χώρα για να δώσει μια βιώσιμη υποστήριξη σε αυτούς που επιστρέφουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα για την επανένταξη. 200 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για το Αφγανιστάν. Όλα αυτά προέρχονται από την αναπτυξιακή βοήθεια. Από ένα ειδικό κεφάλαιο το οποίο έχει ε, το οποίο προορίζεται ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε υπηρεσίες του ΟΗΕ, σε τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε εταίρους που δρούν με βάση το πνεύμα που διέπει και τον ΟΗΕ. Μιλώ για την UNICEF, την ε, πατιαρμοστία για τους πρόσφυγες κλπ. Τώρα, για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Και εμείς γνωρίζουμε τα αποτέλεσματα κάποιων ερευνών που έγιναν από τη Save the Children και από άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσει. Και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να ενημερώσουν για οποιασδήποτε περιπτώσεις ανηλίκων γνωρίζουν που επιστρέφονται στο Αφγανιστάν εκτός της νομικής, εκτός του νομικού πλαισίου που διαθέτουμε για τις επιστροφές. Όλες οι επιστροφές ανηλίκων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας αναφέρουν τα κράτη-μέλη, ε, γίνονται είτε ως τμήμα μιας οικογένειας, δηλαδή επιστρέφει όλη η οικογένεια, είναι εθελοντικές επιστροφές οι οποίες οποίες παρακολουθούνται επαρκώς και ηχνηλατώνται από τα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το τέρμιναλ στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, στο κείμενο της κοινής πορείας των μέλλον πράγματι γίνεται μια αναφορά για ένα τέτοιο τέρμιναλ. Οι αφγανικές αρχές ανησυχούσαν για το γεγονός ότι ενδεχομένω θα ήταν πολύ μεγάλη η αριθμή των επιστρεφόντων ε, επιστρεφωμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό το λόγο και οι αρχές άλλαξαν γνώμη και δεν μας ζήτησαν να τις βοηθήσουμε σε κάτι τέτοιο, στη δημιουργία ενός τέτοιου ιδιαίτερου τέρμιναλ. Οπότε δεν έχουμε και κανένα κονδύλιο εγγεγραμμένο στον προπολογισμό γι' αυτό. Πρόεδρος, πριν απευθεώ στην κυρία Χαμίντη, Σοφή, ήθελες και εσύ να κάνεις ένα ερώτημα σύντομο. Δύο, λέει η κυρία Εντβέλτ. Λέτε ότι λαμβάνετε υπόψη τι εκθέσει των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά τελικά βασίζεστε σε αυτά που σα λένε τα κράτη-μέλη. Παράξενο. Διότι η κυβέρνηση, η δική μου κυβέρνηση, λέει ότι δεν παρακολουθεί τι συμβαίνει σε αυτά τα άτομα όταν επιστρέψουν. Δεύτερον, διαδικαστικό. Σα ρωτήσαμε γιατί η κοινή πορεία για το μέλλον και είπατε με ένα έτσι λίγο κοινικό τρόπο ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό παράξενο, γιατί στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη είναι ε, ένα τμήμα του, της νομοθετικής αρχής, είναι το Συμβούλιο. Ε, εμείς είμαστε το άλλο τμήμα. Όταν εμείς σας ζητάμε κάτι, δεν θεωρείτε ότι πρέπει σόν και καλά να ακολουθήσετε τη συμβουλή μας. Δεν καταλαβαίνω. Πώς βλέπετε το ρόλο σας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει η Κομισιόν ε, απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Ε, είμαι μη πολιτικό μέλος της Κομισιόν και θέλω να παραμείνω στα όρια αυτά. Στη δεύτερη ερώτηση, που είναι πιο πολιτική, θα πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που κάνει είναι να, να δίνει συνέχεια στα αιτήματα και αυτής της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Και σας είπα ότι σας δίνουμε όλες τις πληροφορίες και τη διαφάνεια που μπορούμε σύμφωνα με τους κανόνες και σας ενημερώνουμε για το πώς διαπραγματευόμαστε αυτές τις συμφωνίες. Για το θέμα του, του follow-up, της παρακολούθησης, όλα τα προγράμματα επανένταξης τα οποία ανέφερα διαθέτουν διατάξεις για την παρακολούθηση ε, του πώς γίνονται οι επιστροφές και το τι γίνεται μετά τις επιστροφές. Οπότε ε, έχουμε τέτοιες πληροφορίες τώρα για περιπτώσεις που φύγουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωνία των πολιτών. Ε, πρέπει να βασιστούμε στα κράτη, στις προφήσεις που μας δίνουν τα κράτη-μέλη, γιατί αυτά είναι που υλοποιούν τη Frontex. Οι ίδιες οι πτήσεις επιστροφής παρακολουθούνται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο. Οπότε από τα κράτη-μέλη θα πάρουμε πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μας πιέζει ο χρόνος, αλλά κυρία Χαμίντη, εσείς έχετε το τελευταίο λόγο. Καταλαβαίνετε, ε, βλέπετε ότι το Κοινοβούλιο προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Μπορείτε ενδεχομένως να μας διαλευκάνετε τα πράγματα, να μας διαφωτίσετε. Ευχαριστώ. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τη μοίρα των Αφγανών που επιστρέφουν στη χώρα τους. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία απλώ. Είμαι από το Αφγανιστάν, εργάζομαι εκεί και μιλώ με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τη ζωή τους και την οικογένεια τους και να γυρίσουν στην Ευρώπη. Επιστρέφονται σε μια κατάσταση που πρέπει να ξαναξεκινήσουν από το μηδέν. Αυτό έχει πολύ αρνητικές συνέπειες και στη δική του ζωή και στη ζωή των οικογενειών τους. Και οι, κατά, οι συνθήκες ασφαλείας απαγορεύουν στα παιδιά να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, ε, δυσκολεύονται να βρουν δουλειά οι ίδιοι και ταυτόχρονα ορισμένοι από αυτούς που επιστρέφονται δεν έχουν καν γεννηθεί στο Αφγανιστάν. Οπότε πηγαίνουν σε μια καινούρια χώρα, τελείως ξένη για αυτούς. Με διαφορετικό τρόπο ζωής, κάτι που δυσχεραίνει πολύ περισσότερο την κατάστασή τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις, ε, που μοιράζετε τις ανησυχίες σας μαζί μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη στο Αφγανιστάν. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συσπηρωθούμε για να σώσουμε ζωές ανθρώπων που υφίστανται άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους καθημερινά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που μόλις ε, κάναμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τον έλεγχο μάλλον από κοινού με την Επιτροπή Ανάπτυξης για να βλέπουμε πώς ε, κινείται η δυναμική στο Αφγανιστάν και να μαθαίνουμε τι συμβαίνει ώστε να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. you. Dear colleagues, um, the next item on the agenda is uh, Συνάδελφοι, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι ο διαρθρωμένο διάλογο με τον Επίτροπο, τον κύριο Βερμοπλό. Καλώ ήρθατε. Και μεταξύ των πολλών θεμάτων που έχουμε να συζητήσουμε, ε, είναι προφανή, απλά να αναφέρω μερικά από αυτά. Έχουμε την κατάσταση στη Μεσόγειο, η εφαρμογή του προγράμματο εργασία και οι προτεραιότητες για το 2019. Χαίρομαι που έχει έρθει ο κύριος Επίτροπος ε, και ξέρω πως ε, θέλετε να συζητήσετε μαζί του. Δίνω λοιπόν το λόγο αμέσως και χωρίς χρονοτριβή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλοντ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι. Πίστεψτε με, χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι εδώ. Και βεβαίως ε, πάντα μας ε, βοηθάει αυτός ο διάλογος να δούμε τα διάφορα προβλήματα. Ο διάλογος μας, ε, ειδικά σήμερα, είναι πολύ επικαιρός γιατί θα μας επιτρέψει να ορίσουμε στόχους σε σχέση με την ολοκλήρωση της συνολικής στρατηγικής για τη μετανάστευση και την ασφάλεια η μετανάστευση και η ασφάλεια είναι τομείς όπου η ένωσή μας και η δουλειά που κάνουμε εδώ έχει σαφή προστιθέμενη αξία ε, για τους πολίτες μας. Τα ζητήματα αυτά είναι οι δύο κορυφαίες ανησυχίες τους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε αποτελέσματα στις πρωτοβουλίες μας και για τη μετανάστευση και για την ασφάλεια. Οπωσδήποτε πριν από τις εκλογές και όχι μόνο για να δοθεί αυτή η αίσθηση της ε, προστιθέμενης αξίας, αλλά και με επιχειρησιακά μέτρα να βλέπουν μια διαφορά επιτόπου. Τα συγκεκριμένα παραδοτέα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πολιτική ατμόσφαιρα, το πολιτικό κλίμα της προεκλογικής περίοδου. Σας. Καλό λοιπόν εσάς, την Επιτροπή Λίβε να κάνετε τις εκθέσεις για όλες τις νομοθετικές προτάσεις το αργότερο τον Νοέμβριο. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε συζητήσει με την Προεδρία του Συμβουλίου πριν από τον Ιανουάριο. Όλοι γνωρίζετε ότι ο χρόνος πιέζει. Και είμαι εδώ για να στηρίξω το έργο σας. Να σας δώσω τώρα μια γενική εικόνα των τελευταίων εξελίξεων και προκλήσεων που έχουμε τους μήνες που έρχονται στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας, όπως ξέρετε. Ένα μεγάλο κομμάτι της ομιλίας για την κατάσταση της Ένωσης αφιερώθηκε σε έναν αριθμό σημαντικών νέων προτάσεων που θα ενισχύσουν και θα συμπληρώσουν την δουλειά που κάνουμε σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Θα ξεκινήσω με τα θέματα της μετανάστευσης μέρος της ε, συνολικής στρατηγικής και κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι είναι η σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Άρα προτείναμε να ενισχύσουμε και να εξοπλίσουμε την Ευρωπαϊκή Συνοριακή και Ακτοφυλακή, Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή με ενισχυμένους πόρους και αρμοδιότητες για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη και να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα. Τα προτινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν την σύσταση ενός μόνιμου προσωπικού 10.000 ατόμων μέχρι το 2020 και μια ισχυρότερη εντολής για τις επιστροφές. Η υπηρεσία τώρα θα μπορεί επίσης να κάνει κοινέ επιχειρήσεις και να αναπτύσσει προσωπικό σε όλες τις τρίτες χώρες προτεραιότητας και όχι μόνο στις γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάντα κατόπιν συμφωνίας της Ένωσης με τις Μεταξύ του 2021 και 2027 προτείνουμε να ενισχύσουμε τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας σε ένα σύνολο 11,3 δισεκατομμυρίων. Με αυτόν τον αυξημένο προϋπολογισμό η υπηρεσία θα είναι σε θέση να αποκτήσει δικό του εξοπλισμό, δηλαδή σκάφη, αεροσκάφη και οχήματα και έτσι σταδιακά να ανεξαρτητοποιηθεί από το υλικό των κρατών μελών. Έτσι δεν θα χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε πλέον καταστάσεις όπου η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων θα διακυβεύεται λόγω κενών στον εξοπλισμό. Και έτσι, αν δεν αντιδρούν αρκετά γρήγορα τα κράτη-μέλη ή δεν συνεισφέρουν καθόλου. Ταυτόχρονα προτείνουμε να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου. Η πρόταση της Κομισιόν ακολουθεί το κείμενο το οποίο συμφωνήσατε εσείς προσωρινά με το Συμβούλιο. Η υπηρεσία θα πρέπει να εξοπλιστεί πλήρως για να παρέχει μια γρήγορη και πλήρη στήριξη στα κράτη-μέλη σε όλη αυτή την διαδικασία. Η υπηρεσία θα μπορεί να παρέχει στήριξη στα κράτη-μέλη στην διοικητική διαδικασία για διεθνή προστασία αλλά και για τη διαδικασία του συστήματος του Δουβλίνου. Η ενισχυμένη αυτή υπηρεσία θα συνεργαστεί χέρι-χέρι με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Μαζί θα μπορούν να αναπτύσσουν στήριξη, ομάδες στήριξης διαχείρισης της μετανάστευσης εκεί όπου χρειάζεται. Σε hot spot μεταξύ αυτών και σε κέντρα ελέγχου. Και οι δύο υπηρεσίες επίσης ε, θα συνεργάζονται στις επιστροφές. Έτσι θα υπάρχει καλύτερη συνεργασία και μεταξύ των διαδικασιών επιστροφών και ασύλου. Και όπως είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε κι εσεί μόνο μία πτυχή της μεταναστευτικής μας πολιτικής. Μία άλλη, εξίσου σημαντικό τμήμα μια πτυχη τη μεταναστευτική μα πολιτικης πολιτικής είναι να ενισχύσουμε τις νόμιμες ε, διόδου ε, και για σκοπούς προστασίας αλλά και για τις ανάγκες των οικονομιών μας. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω την πολιτική των επιστροφών, η Κομισιόν πρότεινε μια στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας επιστροφών. Αυτό. Λοιπόν, η διαδικασία αυτή θα δει τις διαδικασίες επιστροφών και θα μειώσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα τη μελη στις επιστροφές, ενώ θα περιέχει και τις απαραίτητες διασφαλίσεις για τους ταυτόχρονα με την αυξημένη στήριξη της ε, συνοριοφυλακής ε, στο θέμα των επιστροφών η συνεργασία με τρίτες χώρες στην επανεισδοχή και η σημαντική οικονομική βοήθεια που θα είναι ε, διαθέσιμη στην ΑΜΥΦ θα συνεισφέρει σε πιο αποτελεσματικές επιστροφές και θα παίξει και ένα ρόλο σε μια βιώσιμη πολιτική μετανάστευσης. Η έγκριση των προτάσεων του Σεπτεμβρίου είναι θέμα προτεραιότητας. Έχει ξεκινήσει ήδη η δουλειά στο Συμβούλιο ή θα ξεκινήσει για όλα αυτά τα θέματα. Οπότε, καλωσορίζω την έγκαιρη έγκριση των εκθέσεων της Επιτροπής σας. Θα γίνει η πρώτη συζήτηση σε βάθος με τους υπουργού Εσωτερικών την Παρασκευή στο Λουξεμβούργο, όπου θα θέσουμε και το θέμα ενός κοινοβεπαϊκού συστήματος ασύλου. Τώρα, να στραφώ στο εξής. Η επίτευξη συμφωνίας ε, σε όλα αυτά τα σημεία είναι πρώτη προτεραιότητα για ένα σύστημα που θα αντέχει στις κρίσεις. Ε, μέρος αυτού του συστήματος είναι η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Μόνο ένα πιο αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα του Δουβλίνου μπορεί να εκφέρει μια πραγματική αλλαγή τώρα και στο μέλλον. Ελπίζω ότι η Αυστριακή Προεδρία θα συνεχίσει να προσπαθεί να επιτύχει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ευθύνη και της αλληλεγγύης και οι διαπραγματεύσεις μαζί σας να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν για το Eurodac, την βάση δεδομένων. Χαιρετίζω την προσωρινή πολιτική συμφωνία. Η κυρία Μακοβέη ε, εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για το θέμα αυτό. Τα εκκρεμή ζητήματα επίσης πρέπει να συμφωνηθούν το συντομότερο δυνατόν. Αυτό είναι σημαντικό και για την διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων. Οπότε θα πρέπει να επιτραπεί να πάμε στην έγκριση του συντομότερο δυνατόν. Για τις τρεις προτάσεις δηλαδή τον ε, κανονισμό της ε, συνθήκες υποδοχής ε, και το συνολικότερο πλαίσιο του Δουβλίνου, χαιρετίζω την προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθη επί Βουλγαρικής Προεδρίας και είμαι πεπισμένος ότι η Αυστριακή Προεδρία θα κάνει λίγες αλλαγές και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε τις συζητήσεις με το Συμβούλιο για να οριστικοποιηθούν σύντομα αυτές οι προτάσεις. Επίσης πρέπει να σημειωθεί πρόοδο στον κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου. Ελπίζουμε το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε μια διαπραγματευτική εντολή για να ξεκινήσει σύντομα ο τριμερής διάλογος. Όπως είπα, πρέπει να σημειωθεί πρόοδο σε όλα τα θέματα της συνολικής προσέγγισης μετανάστευσης και για την νόμιμη μετανάστευση. Ε, η ενίσχυση των νόμιμων διόδων είναι βασικό κομμάτι της μεταναστευτικής μας πολιτικής. Έχει κέρια σημασία να μειωθεί η παράτυπη και ανασφαλής μετανάστευσης και να υπάρχουν ασφαλείς διόδοι για όσους χρειάζονται προστασία και να υπάρχει και μια ελεγχόμενη δίωδος για τη μετανάστευση εργασίας θα συζητήσω την πρόταση της μπλε κάρτας με τους υπουργούς της 12 Οκτωβρίου και υπογραμμίζω την σημασία του να συμφωνήσουμε σε μια μεταρρυθμισμένη καινούρια μπλε κάρτα σε... η οποία θα έχει προσθέμενη αξία σε σχέση με την υφιστάμενη. Θα τους παρακινήσω επίσης να προχωρήσουν ε, και να υπάρξουν κάποια πιλωτικά σχέδια νόμιμης μετανάστευσης με επιλεγμένες αφρικανικές χώρες πριν από το τέλος του έτους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και για τις συμφωνίες επανεισδοχής με κάποιες από αυτές, εάν ε, θέλουμε πραγματικά να είμαστε αξιόπιστοι και να έχουμε την πλήρη στήριξη των αρχών των αφρικανικών χωρών στην πρόληψη της ε, παράτυπης μετανάστευσης πρέπει να επεκτείνουμε της ευκαιρίας νόμιμης μετανάστευσης ή τουλάχιστον να είναι ευκολότερο να υπάρχει πρόσβαση στις υφιστάμενες διόδους. Τέλος, θα ζητήσω από τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ε, τις υποσχέσεις τους περί μέντε κατάστασης και να προχωρήσουν οι συζητήσεις για ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο των συντομότερων δυνατών. Να αναφέρω τώρα και τις ε, προτάσεις ε, της Κομισιόν του Μαρτίου. Ο στόχος ε, της πρότασης είναι να γίνει ευκολότερο και γρηγορότερο το να βγάζουν οι ταξιδιώτες βίζα, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθούν οι έλεγχοι ασφαλείας. Επίσης, στηρίζει και την πολιτική επιστροφών, τονίζοντας την σημασία της συνεργασίας των τρίτων χωρών για την επανεισδοχή παρατύπων μεταναστών. Έχουμε προτείνει αυστηρότερους κανόνες ε, για την επεξεργασία χωρών ε, αιτήσεων από τις χώρες που δεν δέχονται επαρκώς ε, τις επιστροφές με έναν μηχανισμό διαφανή και στοχευμένο. Η Προεδρία ήδη έχει μια διαπραγματευτική εντολή, οπότε ελπίζω η ΛΥΜΠΕ επίσης προσεχώς να εγκρίνει μια σχετική έκθεση. και πάλι για τα ζητήματα της ΒΙΖΑΣΗ Κομισιόν θα συζητήσει τα ζητήματα αυτά της αμοιβαιότητας με τις ΗΠΑ και τον Καναδά και θα, τα, σας ενημερώσω ξανά. Ξέρω πως παρακολουθείτε στενά το θέμα. Ανησυχώ και εγώ όσο και εσείς. Γι' αυτό θέλω να επαναλάβω την πλήρη μου δέσμευση για να σημειωθεί συγκεκριμένη πρόοδος για την πλήρη αμοιβαιότητα βίζας με τη ΣΥΠΑ έθεσα αυτό το ζήτημα και το θέτω σε κάθε ευκαιρία. Θα πάω στην Ουάσιγκτον τον επόμενο μήνα και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Θέλω να είμαι σαφής και κατηγορηματικός ως προς αυτό. Οι τεχνικές επαφές συνεχίζονται. Και όπως είπα θα συνεχίσω τις συζητήσεις το πολιτικό κλίμα στην Ουάσιγκτον δεν μας ευνοεί, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αμοιβαιότητα στην βίζα για τα κράτη-μέλη μας. Η Κομισιόν, και όπως ξέρετε αυτό με απασχολεί προσωπικά, έχει στόχο ακριβώς να διατηρήσει την ζώνη Σέγγεν. Το λέω ξανά και θέλω να είμαι σαφής. Προσωρινή εσωτερική έλεγχη στα σύνορα δεν πρέπει να γίνουν μόνιμοι. Άρα είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε και στο ποια είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας μετακίνησης αφενός ε, και της ασφάλειας αφετέρου. Για τον λόγο αυτό έχουμε προτείνει την τροποποίηση του κώδικα Σέγγεν όχι για να απαντήσουμε σε τρέχουσες πρακτικές. Και πάλι ελπίζω η Λίμπε να εγκρίνει την έκθεσή της για να ξεκινήσουν τριμερείς διάλογοι πριν από το τέλος του έτους. Η Προεδρία έχει ήδη εντολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέους κανόνες για να μην υπάρχουν καταχρήσεις και να ακολουθούν όλοι τους κανόνες. Αγαπητοί φίλοι, να αναφερθώ τώρα στα θέματα ασφαλείας, όπου με την δική σας την συνεισφορά γίνονται μεγάλες προσπάθειες για μια αποτελεσματική ένωση ασφαλείας. Έχουμε λοιπόν μια ολοκληρωτική αλλαγή παραδείγματος όσον αφορά την συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στην Ευρώπη. Ξεπερνάμε παλιά ταμπού που έλεγαν ότι η ασφάλεια είναι προνόμιο των κρατών μελών. Αντιμετωπίζουμε πολλές ε, απειλές. Η αντιμετώπιση τους όμως ε, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και ένας κοινός στόχος. Το γεγονός ότι δεν είχαμε εδώ και ένα χρόνο μια μεγάλη τρομοκρατική επίθεση από τη Βαρκελόνη τον Αύγουστο πέρσι, ίσως δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Παρουσιάσαμε ένα σημαντικό σχέδιο κανονισμού για την πρόληψη διάδοσης τρομοκρατικού υλικού στο διαδίκτυο. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν ως απάντηση στις εκκλήσεις Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να ενισχυθούν τα μέτρα για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδικτύο. Αυτό επίσης βασίζεται και στην πρόοδο που είχε σημειωθεί στο σχετικό φόρουμ για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και ενώ σημειώνεται αυτή η πρόοδος όσοι σχεδιάζουν τρομοκρατικά χτυπήματα εξακολουθούν να διασπείρουν την δηλητηριώδη προπαγάνδα του στο διαδίκτυο με σχετική ευκολία. Είναι σαφές ότι πολλές από τις εταιρείες οι οποίες ακολουθούν την εθελοντική προσέγγιση έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να μην υπάρχει εκμετάλλευση των πλατφορμών από τρομοκράτες. Επίσης είναι αλήθεια ότι πολλές εταιρείες δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Μια σειρά δικλείδων ασφαλείας ε, επίσης ε, περιέχονται στον κανονισμό για να μην υπάρχει αφαίρεση αθώου περιεχομένου και να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τζούλιαν Κίνγκ επίσης θα σας δώσει κάποιες λεπτομέρειες αργότερα σήμερα. Η ριζοσπαστικοποίηση επιτόπου, εκτός διαδικτύου, είναι εξίσου σημαντική. Και εκεί πέρα λοιπόν εργαζόμαστε εντατικά για να υπάρχει κάποια ακτή, απτή προσθέμενη αξία στα κράτη-μέλη και στους ανθρώπους που εργάζονται πάνω στο θέμα. Η σύσταση της ομάδας, ε, της κατευθυντήριας για το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης είναι το πρώτο ορόσημο που υπάρχει στην, στο μέτωπο της πρόληψης. Τώρα να αναφέρω μια άλλη σημαντική προτεραιότητα η διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων μετανάστευση συνόρων και ασφάλειας. Συναδελφοί, είναι ευθύνη μα να καταστήσουμε πραγματικότητα τη διαλειτουργικότητα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε του πολίτε μα. Εκτιμώ την εργασία και τι προσπάθειε που έχουν καταβάλει οι εισηγητέ Λάνερ και Μέλο, καθώ και οι Σκιώδη, ώστε να βρουν συμβιβαστικέ τροπολογίε και να εγκρίνουν την έκθεση, υιοθετήσουν την έκθεση του την επόμενη εβδομάδα. Η Προεδρία ήδη έχει εντολή για διαπραγμάτευση και προσβλέπω στην έναρξη των τριμερών διαλόγων. Έχουμε επίσης ε, πιτάπετος ε, τη ΕΕΣ μεγάλη πρόκληση αλλά με πολύ πεπειραμένους εμπειρογνώμονες. Επίσης, όσον αφορά το ίδιο Λίζα, επίσης ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακοβέη και τους Κιώδης για την εργασία τους και για αυτό το θέμα και με χαρά βλέπω ότι ο νέος κανονισμός θα μπει σε εφαρμογή πριν το πέρας του έτους να ευχαριστήσω με την ευκαιρία όλους σας για όλη σας την εργασία για το ετίας, το, το σύστημα εισόδου-εξόδου και την μεταρρύθμιση Σέγγεν 2. Η έγκριση αυτών των προτάσεων θα ενισχύσει την ιστορική ασφάλεια, θα διευκολύνει τη διέλευση και θα βοηθήσει να περιχαρακωθεί η πολιτική της Ένωσης για απελευθέρωση των θεωρήσεων. Να τονίσω δε ε, ε, ακόμη περισσότερο ότι η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι προαπαιτούμενο για τη σωστή λειτουργία του Σέγγεν και την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σέγγεν. Επίσης, ε, προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας για τις προτάσεις για πρόσβαση στις οικονομικές πληροφορίες διασυνοριακά, δηλαδή πρόσβαση σε ηλεκτρονικές αποδείξεις και αυτό το σύνολο μέτρων που περιλαμβάνει και μια σύσταση για βελτίωση των ελέγχων και την ανιχνευσιμότητα ε, των ε, όπλων θα βοηθήσει στον περιορισμό των δρομοκρατών και του χώρου δράσης τους. Ελπίζω λοιπόν πως θα έχουμε εκθέσεις εδώ, ώστε να τις εκθέσεις που θα εγκριθούν σύντομα, ώστε να ξεκινήσουν οι τριμερείς όσο γίνεται πιο σύντομα. Επίσης, ε, προσβλέπω στη συνεργασία με την κυρία Κάουφμαν, ώστε να εξασφαλίσουμε μια ομαλή έγκριση της πρότασης για την καταπολέμηση της απάτης μη μετρητών, για να προστατευτούν καλύτερα οι πολίτες ενάντια σε αυτά τα ε, αδικήματα καθώς και να βελτιώσουμε την ε, προστασία και την δυνατότητα επιβολής του νόμου. Τέλος, δύο λόγια για τη χρηματοδότηση. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα εξακολουθήσουν να παίζουν κρίσιμο ρόλο για την επίτευξη των στόχων και φιλοδοξιών σε όλους τους τομείς πολιτικής μια ενδιάμεση αξιολόγηση της, ε, των κονδυλίων για μετανάστευση και την ασφάλεια επιβεβαίωσαν την ορθότητα αυτών και την πρόοδο της εφαρμογής τους, της εκτέλεσης τους. Όπως ξέρετε, στον τομέα της μετανάστευσης των συνόρων και της ασφάλειας, η Κομισιόν έχει υποβάλει φιλόδοξη πρόταση στο νέο PDP όπου αντικατοπτρίζεται η μεγάλη προτεραιότητα που δίνουμε για την αντιμετώπιση των μελλοντικών χρηματοδοτικών προκλήσεων. Είναι πολιτικό σημαντικό να τονιστούν οι προσπάθειες για τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και την ασφάλεια με επαρκή ε, χρηματοδότηση, ευελιξία και ένα σύστημα ατολατικτενό έλεγχο για την πραγματική ε, ε, Υλοποίηση. Επίσης πρέπει να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των μέλωσων που λειτουργούν στην Ένωση αλλά και στις τρίτες χώρες πάντοτε σύμφωνα με τους στόχους των πολιτικών μας. Η Κομισιόν υπολογίζει στο Κοινοβούλιο, βασίζεται στο Κοινοβούλιο για τη στήριξη των προτάσεών της, για την ομαλή διαπραγμάτευση και για την συνεργασία με το Συμβούλιο για έγκαιρη υιοθέτηση αυτών. Γνωρίζω πως ήδη έχετε αρχίσει την εξέταση των νέων νομοθετικών προτάσεων και τώρα είναι ο καιρός να προχωρήσουμε ε, στιάζοντας ε, ε, στα θέματα και αντιμετωπίζοντας τα. Εγώ προσωπικά και οι υπηρεσίες μου προσβλέπουμε στη συνεργασία με την Επιτροπή σας και βεβαίως όλος ιδιαίτερος με τους εισηγητές Φαγιόν, Χολμάγερ, Λένερς και Ντέλη. Αγαπητοί φίλοι, όλοι γνωρίζουμε πως έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και ότι ο χρόνος που έχουμε στη διαθεσή μας είναι περιορισμένος. Ανατρέχοντας την πρώτη μας συνεδρίαση, τη δική μου ακρόαση πριν από τέσσερα χρόνια, βλέπω πως έχουμε επιτύχει πολλά μαζί. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι πως έχουμε ε, συνεργαστεί ε, ικανοποιητικά όλα αυτά τα χρόνια. Εάν θυμάμαι καλά, μου, είπατε, μου είπανε οι συνάδελφοι πως έχει να αντιμετωπίσει την πιο δύσκολη επιτροπή. Τέσσερα χρόνια μετά όμως θα πρέπει να σας πω ότι ποτέ στη ζωή μου δεν είχα τόσο επικοδομητικές σχέσεις με βουλευτές. Σα ευχαριστώ γι' αυτό. Έχουμε ακόμα 8 μήνες στενή συνεργασία και προσήλωση για να μπορέσουμε, όπως έλεγα, να ολοκληρώσουμε τις στρατηγικές μας. Συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει μια μαγική λύση ούτε για το θέμα της ασφάλειας, ούτε για την ε, διαχείριση των μεταναστευτικών Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Θα χρειαζόμαστε να συμφωνήσουμε σε όλα τα ζητήματα της ε, Ένωσης Ασφάλειας και αλληλεγγύη ώστε να έχουμε αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη στις πολιτικές μας. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκής κλίμακας πολιτικές και είμαι βέβαιος ότι οι 8 μήνες που μας περιμένουν θα είναι επικοδομητικοί και αποτελεσματικοί και προσβλέπω στη στενή συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Παρατηρώ ότι συνάδελφοι καθώς μιλούσατε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κουρασμένοι κάποιοι συνάδελφοι, εγώ πάντως πιστεύω ότι αυτά που αναφέρατε σήμερα δεν είναι μόνο φόρτος της Επιτροπής, είναι και δικός μας, το δικό μας έργο. Είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Επίσης θεωρώ πως ε, είναι και δουλειά μας ε, που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της θητείας. Κάθε λοιπόν θέμα είναι σοβαρό, είναι φορτωμένο με πολλά ζητήματα επιμέρους και το βλέπω αυτό στα πρόσωπα των συναδέλφων. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν ζητήσει γι' αυτό το λόγο, όλοι έχουν γραφτεί στον κατάλογο μιλητών. Αυτό που θέλουμε να προσπαθήσουμε είναι να σας ενημερώσουμε σαφώς για το τι ε, πιστεύουμε, γιατί το Κοινοβούλιο έχει κινηθεί πολύ γρήγορα και έχουμε ενημερώσει και το Συμβούλιο. Δεν θα πρέπει λοιπόν κανείς να πει ότι δεν κινούμαστε γρήγορα και θα είναι καλό να καταγραφούν οι απαντήσεις, η αντιπόκριση μάλλον στο αυτό που είπατε για το αν προχωρούμε αρκετά γρήγορα, για το άσυλο, τη μετανάστευση, τα σύνορα. Να καταγραφεί λοιπόν ήδη ότι για τη δέσμη των ε, συνόρων έχουμε βάλει την ε, εισηγήτρια την κυρία ε, Τίλη, την κυρία Σαργεντίνη για την για το ιδέσμι για τις επιστροφές. Υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα, διαλειτουργικότητα ψηφίζεται τη Δευτέρα βεβαίως και πάλι δύσκολο θέμα αλλά ε, εάν δεν τα καταφέρουμε θα πάμε στο στριμερίς. Η κυρία Στίβενς είναι ε, η συγγήτρια για το παράνομο υλικό περιεχόμενο ε, στο online. Ένα σωρό ζητήματα. Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουμε κάθε ένα από αυτά τα θέματα, γιατί το καθένα από αυτά είναι δύσκολο. Ας πούμε για την ε, αμοιβαιότητα θεωρήσεων, είναι καλό αυτό που είπατε, αλλά χρειάζεται λύση. Που να είναι μόνο μία εγκύκλιος ή μια, που να δημιουργεί μια κυκλική κατάσταση. Και για τους Αμερικανούς ε, φίλους μας, έχουμε πάει και εμείς στη Washington, δεν άρκεσε χρειάζεται να κάνουμε μια προσπάθεια περισσότερη πριν το τέλος της, ε, της θητείας και για το Δουβλίνο και για το αδιέξοδο για τη δέσμη για το άσυλο. Εγώ αυτό που βλέπω στο Συμβούλιο είναι το θέμα της ειδικής φιλοψηφίας και της συνένεσης. Εάν η Κομισιόν ε, συνεχίσει με το θέμα της συνένεσης και δεν δεν βλέπω ποια θα είναι η διέξοδο. Δηλαδή μπορεί εμεί να δουλεύουμε για κομμάτια του, Δέσμη δέσμης για το άσυλο, αλλά έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι νομίζετε εσείς. Τι στόχο έχετε, θα το αφήσετε να συνεχίσετε. Το καταλαβαίνω το γιατί, αλλά θα επιμείνουμε με τον κανόνα της, της ομοφωνίας. Γιατί για μένα αυτό ε, ε, ε, δεν οδηγεί πουθενά. Ποτέ δεν πρόκειται να ξεμπλέξει το θέμα του ασύλου. Και έπειτα, δεν ξέρω αν θυμάστε τις ε, διατάξεις ε, σχετικά με αυτό, γιατί δεν βλέπω να σημειώνεται πρόοδο. Πρέπει να το συζητήσουμε, νομίζω. Όσο και αν προσπαθήσουμε εμείς και ακόμα και με υπό την Ρουμανική Προεδρία. Ε, είναι δύσκολο το ερώτημα, αλλά πρέπει να τεθεί. Ας προχωρήσω λοιπόν στον κατάλογο των ομιλητών. Συνάδελφοι, ε, μη μου θυμώσετε, θα ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές ή τους αντικαταστάτες των συντονιστών. Η κυρία συντονιστων κυρια λείπει για το έλκα, αλλά από κατάλαβα ο κύριος Έγγελς θα μιλήσει εξ ονοματός της. Όλοι λοιπόν δύο λεπτά Εάν κάτι δεν έχω καταλάβει καλά, απλά πείτε το μου για να συνεχίσουμε. Δύο λεπτά για να μιλήσετε όλοι. Παρακαλώ να μείνετε στα δύο λεπτά. Πρώτα οι συντονιστέ και μετά θα ζητήσω από τον Επίτροπο να απαντήσει. Φρανκ, πρώτος εσύ από το ΕΛΚ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Κλοντ. Και πήρα και προαγωγή, δεν το περίμενα ερχόμενος εδώ σήμερα και σε κάθε περίπτωση αυτά που θα πω δεν αντιστοιχούν σε αυτά που θα έλεγε κανονικά ένας ε, συντονιστής του ΕΛΚ. Δύο στοιχεία θέλω να σχολιάσω της μεταναστευτικής πολιτικής. Η Κομισιόν ολοκληρώνει την θητεία της όπως και Και ίσως ε, έχει έρθει η στιγμή να δείξει ένα θάρρος το οποίο δεν είχε δείξει στο παρελθόν. Το έχω πει και στον πρόεδρο της Κομισιόν νομίζω ότι και ο ίδιος θα ήθελε να προχωρήσουμε σε θέματα τα οποία έχουν ε, λίγο ε, αδρανήσει. Για το Δουβλίνο καταρχήν να σας πω. Όλοι γνωρίζουμε για το Δουβλίνο ότι το σύστημα επινοήθηκε χωρίς πίεση. Χωρίς μεταναστευτικές πιέσεις. Κάποια στιγμή που ήμασταν άνετοι να επινοήσουμε ένα σύστημα ε, επιμερισμού ε, χωρίς πίεση. Τώρα έχουμε πίεση και υποπίεση αυτό το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα κατανομής μεταξύ όλων. Θα πρέπει να γίνει κατανομή μεταξύ αυτών που το επιθυμούν, που το αντέχουν και που θέλουν να δείξουν ότι υπάρχει αλληλεγγύη σε ένα τμήμα τουλάχιστον της Ευρώπης. Μετά, η επίσημη, η νόμιμη μετανάστευση. Ο Κλοντ και οι άλλοι που ασχολούνται με την ασυνή ε, κάρτα, ε, έχουμε δει ότι η πρόοδος είναι πολύ μικρή. Και τα νούμερα είναι τόσο μικρά που δεν αξίζει να τα, να τα συζητάμε. η νόμιμη μετανάστευση είναι απαραίτητο να οργανωθεί παρόλο που είναι δύσκολο. Γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τους, ε, τις αιτίες, τους ε, λόγους της, ε, που δημιουργούν τη μετανάστευση, αλλά δεν θα τα καταφέρουμε τελικά. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να υποδεχτούμε μεγάλους αριθμούς μεταναστών. Και υπάρχουν κράτη τα οποία είναι έτοιμα κάποια πρόθυμα και άλλα όχι. Και καλύτερο είναι να μην πιεστούν αυτοί που δεν θέλουν, διότι θα ήταν επικίνδυνο και για τους ίδιους τους μετανάστες. Αλλά θα πρέπει ο νομοθέτης να δώσει μια ποσότητα ανθρώπων που θα πρέπει να ενταχθούν και να γίνουν δεκτά, να υποδεχτούμε στην Ευρώπη έτσι ώστε να αποφύγουμε τους παράτυπους μετανάστες. Ευχαριστώ. Ε, ο κ. Έγγελς δεν έχει εμπειρία να συντονιστεί, οπότε μίλησε λίγο παραπάνω. Παρακαλώ πολύ, περιοριστείτε στα δύο λεπτά. Να πω στον Επίτροπο ότι ο Επίτροπος πιέζει το θέμα της μπλε κάρτας στο Συμβούλιο. Είναι δικό μου ε, θέμα και της κυρίας Πινέλη και <laughs> το Συμβούλιο δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όμως ο Επίτροπος πιέζει γιατί από τη μια μεριά κάποιοι υποκρίνονται ότι υπάρχουν νόμιμοι δρόμοι μετανάστευσης ε, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν και ο Επίτροπος πραγματικά προσπαθεί να πολεμήσει εναντίον αυτής της υποκρισίας. Τώρα, κύριε Ζίπελ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας ε, αυτήν την παρουσίαση κάπου χάνω την υπομονή μου και επικραίνομαι. Λέτε κύριε Βραμοπούλη ότι πρέπει να προστατευτεί ο χώρος Σέγγεν, αλλά αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι με κάθε πρόταση της Κομισιόν τρέχεται πίσω από το Συμβούλιο και παρατείνονται οι συνοριακοί έλεγχοι. Δεν προστατεύεται έτσι η Αμοιβαιότητα βίζα. Δεν ξέρω πόσο καιρό το περιμένουμε και λέτε ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε. Ε, φοβάμαι ότι δεν θα το δούμε ούτε σε άλλα πέντε χρόνια. Αν ήμουν η Αμερικανική κυβέρνηση θα γέλαγα. Γιατί πάμε, μας λένε δεν θα κάνουμε τίποτα και εμείς λέμε ναι, ναι, να διαπραγματευτούμε. Ε, δεν μας παίρνουν σοβαρά. Διαλειτουργικότητα. Οπωσδήποτε πάρα πολύ σημαντικό για την ασφαλή. Κύριε Αβραμόπλε, αρχικά η ιδέα ήταν να συνδέσουμε διάφορες βάσεις δεδομένων με τρόπο έξυπνο. Το δέχτηκαν όλοι. Τώρα ακούμε ότι θα φτιάξουμε μια νέα τεράστια βάση δεδομένων με εκατομμύρια άτομα. Κατηγορούμενους, υπόπτους, ε, ταξιδιώτες, ε, θύματα, όλα μαζί. Δεν ξέρω πώς θα ενισχύσει αυτό την ασφάλεια όταν μπουν όλα αυτά σε μια βάση δεδομένων. Τα σύνορα ε, πρέπει να προστατευτούν. Εγώ θα προτιμούσα να λέμε ε, θα πρέπει να προστατευτούν οι άνθρωποι. Εντάξει, αλλά δεκτό και αυτό που λέτε. Τώρα Πώ θα γίνει όμως, ε, έχουμε αποφασίσει μια ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή, η οποία δεν λειτουργεί γιατί τα κράτη-μέλη δεν δίνουν αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί. Παρ' όλα αυτά, ε, κάνουμε τώρα κάτι ε, παραπάνω, δεν ξέρω από πού θα έρθουν αυτά τα λεφτά. Λέτε ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στις επιστροφές. Ναι, οι επιστροφές ήταν πάντα κομμάτι του συστήματος ασύλου δηλαδή να στέλνουμε πίσω στη χώρα προέλευσης αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, αλλά τότε γιατί υπογράψαμε αυτήν την κοινή πορεία για το μέλλον με το Αφγανιστάν και όχι με τις χώρες εκείνες, οι πολίτες των οποίων δεν λαμβάνουν ε, άσυλο. Και επίσης δεν ετέθη καθόλου το ζήτημα της ε, κατάστασης των προσφύγων, ειδικά στην Ελλάδα, στη Μόρια ακούσαμε πράγματα ότι δεν υπάρχει απλά επιβάρυνση, ξεχυλίζουν εκεί πέρα οι εγκαταστάσεις, επιπλέον υπάρχουν κατηγορίες περί διαφθοράς, ότι δεν φτάνουν τα λεφτά στους ε, πρόσφυγες, αλλά κάπου στο δρόμο χάνονται ε, και γι' αυτά θα ήθελα να ακούσω κάποια πράγματα και τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν για αυτές τις κατηγορίες. Για το ECR, κ. Διορέκ, δεν πιστεύετε ότι η ανακοίνωση δημιουργίας νόμιμης όδου για τη μετανάστευση που γίνεται τόσο συχνά εκ μέρου σας ενθαρρύνει την παράτυπη μετανάστευση. Γιατί αδιάκοπα βλέπουμε να αυξάνονται οι αριθμοί των μεταναστών στην Ευρώπη οι μισοί από αυτού έρχονται από το Μαρόκο αυτή τη στιγμή. Τι μέτρα έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να έρθει σε επαφή με τις μαροκινές αρχές για να μετριαστεί αυτή η κατάσταση. Το Μαρόκο δεν είναι Λιβύη, είναι μια σταθερή μοναρχία, μάλλον φιλοδυτική, κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα δύσκολο το Μαρόκο να μπει σε, μια, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης. Τρίτη ερώτηση. Ποιος είναι ο οριστικός απολογισμός σας για τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργασίας στον τομέα της μετανάστευσης. Δεν μιλώ τόσο πολύ για τα μέτρα που λάβατε, αλλά για την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι η κατάσταση της Ευρώπης στον τομέα της μετανάστευσης είναι καλύτερη από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια, το 2014. Ευχαριστώ. Thank you. And, uh, for um, uh, Natalie, please. Η Νάταλη για τους φιλελεύθερους. Α, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Ε, μπερδεύτηκα. Ε, Νατάλη, έχεις δίκιο. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την παρουσία του και για την αποφασιστικότητά του. Και ό,τι φορά τα όσα είπε ο Κλοντ, συμφωνώ με τις ερωτήσεις του όσα υπογράμμισε για το θέμα της ε, συνένεσης και της ομοφωνίας, για παράδειγμα. Ε, έχουμε βαλτώσει. Ευχαριστώ επίσης τον Επίτροπο για την υπόμονή του, γιατί πράγματι είναι απογοητευτικό να βλέπουμε αυτή την παράλυση σε πολλά θέματα, όπως για παράδειγμα αυτό της μπλε κάρτας, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, ένα αριθμό υποκριτών. Σε ό,τι αφορά τα όσα μας είπατε, κύριε Επιτροπέ, θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριος για την βελτίωση των συνθήκων υποδοχής των ε, προσφύγων. Ο κ. Αντού σήμερα ε, μας, ε, από την ΕΑΣΟ μας μίλησε για μια μείωση των ετούντων άσυλο, η οποία ξεκίνησε από το 2017 γύρω στο 40% σε σχέση με το 2016, μείωση η οποία επιβεβαιώνεται και μέσα στο 2018. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση στα σύνορα εξακολουθεί να είναι ανησυχητική, ιδιαίτερα ε, στα hot spot της Ελλάδας. Ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων ε, δεν είναι απόλυτα σαφής, αλλά είναι πολύ ψηλός. Επίσης καταγγέλλονται σημαντικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Παραβιάσεις οι οποίες λέγεται ότι επηρεάζουν ιδιαίτερους τους πιο ευάλωτους, δηλαδή τα παιδιά τα οποία ζουν σε δραματικές συνθήκες. Και ανθρωπιστικά και πολιτικά. Στο Ξυμβούλιο από την άλλη μεριά οι οποιασδήποτε μεταρρυθμίσεις έχουν μπλοκαριστεί. Οπότε, κατά την άποψή σας, τι περιθώριο ελιγμών έχετε μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Πολλές φορές έχετε πει ότι είστε αισιόδοξο. <laughs> τι, περιθώριο λοιπόν έχετε. Okay, um, Ο κ. Μωράης για την Γκουε, η Μπάρβαρα Σπινέλη. Συγγνώμη, ξέχασα τους πράσινους. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει σήμερα. Η Γιούντιθ είναι η συντονίστρια των Πρασίνων. Γιούντιθ, έχει το λόγο. Και, πρωτη... και αντιπρόεδρος. Ακούγοντας τον κύριο Αβραμόπουλο, άκουσα πολλές φορές ότι ελπίζει πως θα ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος πριν τις εκλογές. Το είπε πολλές φορές, δεν ξέρω πόσες δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε εκεί και δεν είμαι σίγουρη αν θα έπρεπε κιόλα. Γιατί πολλοί από τους φακέλους ε, δεν έχουν καθυστερήσει εξαιτία ημών, αλλά εξαιτία του Συμβουλίου. Λέει ο Επίτροπος ότι χαίρεται που βλέπει πως υπό την Βλυγουλιαρική Προεδρία καταλήξαμε σε κάποιες προς πρώτες συμφωνίες, προκαταρκτικές συμφωνίες και ότι η Αυστριακή Προεδρία τι είπε, θα κάνει κάποιες πρόσθετες αλλαγές, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Μιλήσατε με επενδυτικά λόγια για την κυρία Μακοβέη, αλλά και εγώ να μιλήσω και για την κυρία Μπιόρκ που δεν είναι εδώ σήμερα από την ΚΟΕ, που πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο για την επανεκατάσταση. Τώρα το Συμβούλιο θέλει πρόσθετες αλλαγές, δεν είναι πρόσθετες. Ή υπάρχει συμφωνία, αυτή που στην οποία καταλήξαμε ή δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις επί αυτών των συμφωνίων. Δεν γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προασπίζουμε την ενότητα των νομοθετικών κειμένων και της διαδικασίας. Και ενώ το Συμβούλιο σπαταλάει το χρόνο του να μιλάει για τις ε, πλατφόρμες αποβίβασης και δεν ξέρω και τι άλλο θα επινοήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Και αν δεν σταματήσουν να το κάνουν αυτό, να ασχοληθούν σοβαρά με τα θέματα, δεν θα δούμε πρόοδο. Είπατε και για τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Για την προστασία των ατόμων και για τις ανάγκες της οικονομίας μας είπατε. Τι ακριβώς εννοείτε. Οι, νόμ, οι οδοί δεν υπάρχουν μόνο για αυτά τα δύο πράγματα, την προστασία των ατόμων και για την οικονομία μας, αλλά και για να εξασφαλίσουμε μια συνεργασία, δίκαιη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Προσπαθούμε να υπογράψουμε συμφωνίες επανεισδοκής και αυτό εξαιτία του ότι δεν υπάρχουν νόμιμες οδοί μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι, νομικές, οι νόμες αυτές οδοί δεν πρέπει να είναι η μετεγκατάσταση. Ευχαριστώ. Μπάρμπαρα Σπινέλη για την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα εστιάσω στην μετανάστευση και ιδιαίτερα σε ορισμένα σημεία επί των οποίων θα ήθελα να έχω απαντήσεις από πλευρά σας κύριε Επίτροπε. Πρώτο, το σύστημα των hot spot. Μόνο το 2018 στην Ελλάδα 18.500 μετανάστες ε, μεταφέρθηκαν από τα νησιά στην ε, υπηρετική Ελλάδα και η κατάσταση δεν βελτιώνεται γιατί τα hot spot αμέσως ξαναγεμίζουν πέραν κάθε ε, δυνατότητας και άρα λοιπόν η ερώτησή μου είναι, δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρηθεί το σύστημα των hotspot, νόμι μεσοδή. Διερωτώ με αν αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε να μιλάμε για πράγματα που δεν υπάρχουν και που το Συμβούλιο αρνείται. Μπλε κάρτα. Για την μπλε κάρτα ήδη πόθηκαν όλα από τον εισηγητή Κλοντ Μωράες. Και αυτό που εγώ θέλω να σας ρωτήσω είναι μήπως θα έπρεπε να καταγγέλουμε τον την αντίσταση του Συμβουλίου και ιδιαίτερα του κανόνα της ε, συνένεσης, γιατί ποτέ δεν πρόκειται να βρεθεί συμφωνία για οποιαδήποτε φάκελο της δέσμες για το άσυλο, αν συνεχίσουμε ε, κατά αυτόν τον τρόπο. Νόμεμη οδός, ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Ε, σήμερα η Επιτροπή μας υπερψήφισε αυτού του είδους της θεωρήσεις. Θέλω να ξέρω τι θα κάνει η Κομισιόν. Άλλο σημείο είναι οι πολιτικές κλεισίματος λιμανιών και συνόρων στην Ιταλία. Και δικαίως επικρίνονται. Αυτό που σας ρωτώ είναι... Αυτό δεν είναι η μοιραία συνέπεια της εξωτερικευσής που αποφασίστηκε από τα κρατημέλη και από την Κομισιόν και της αποτυχίας της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου και εδώ επαναρχόμαστε στο θέμα του συνένεσης και του αδιέξοδου στο Συμβούλιο. Και τέλος, Frontex. Μία μόνο ερώτηση. Νομίζω πως η πρόταση μεταρρύθμισης δεν περιλαμβάνει ενίσχυση της εντολής του Search and Rescue, έρευνα και διάσωση. Και λοιπόν τότε ποιος πια θα μείνει να κάνει έρευνα και διάσωση αφού τα σκάφη των ΜΚΟ πλέον unblock θεωρούνται εγκληματίες. thank you very much, Σας ευχαριστούμε. Η Τζούντιθ ε, ανέφερε την κυρία Μπιόρκ που προφανώς είναι η συγγήτρια για το θέμα να ρωτήσω εξ ονοματός της είχε θέσει το θέμα πότε δηλαδή η Κομισιόν σκοπεύει να υποβάλει την πρόταση αυτή για τα διάθετα κονδύλια για τις ε, μετεκαταστάσεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε σήμερα ή κάποια άλλη στιγμή. Αυτοί ήταν οι συντονιστές συνάδελφοι και έχουμε 8 συνάδελφους θέλουν το λόγο. Υπάρχει κάποιος ε, που δεν έχει ζητήσει λόγο Σόφη. Θες να μιλήσεις. Ε, ναι. Οπότε... Τώρα. Θα απαντήσετε τώρα στους συντονιστές και μετά να ακούσουμε τους υπόλοιπους βουλευτές. Ό,τι θέλετε. Ναι, ναι, και εσείς. Αλλά μπορείτε να είστε λογικά σύντομος ε, και μην τα απαντήσετε όλα. Τώρα έχουμε και άλλους συνάδελφους. Ε, ξέρετε, εμένα μου αρέσουν οι προκλήσεις λέει ο κ. και σημείωσα τις παρατηρήσεις εδώ των συναδέλφων. Είπατε, κάποιος είπε ότι μετά από τέσσερα χρόνια κοινών προσπαθειών, μπορώ να σου πω, είμαστε όλοι κουρασμένοι, αλλά είμαστε και γεμάτοι ενέργεια και αποφασιστικότητα για να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας. Έχουμε 8 μήνες μπροστά μας και όπως είπα στην αρχή βασίζομαι στην συνεργασία σας γιατί ό,τι έχουμε πετύχει βασίζεται σε αυτήν την συνεργασία εάν το Συμβούλιο ήταν σε θέση να ακολουθήσει το αριθμό του Κοινοβουλίου η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη αλλά είμαστε εδώ ακριβώς για να ανανεωθεί το πνεύμα της συνεργασίας και να επαναλάβουμε την αποφασιστικότητά μας για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο. Να οριστικοποιήσουμε δηλαδή αυτά τα οποία έχουμε ξεκινήσει. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις στρατηγικές. Κλοντ. Ευχαριστώ να γίνει μια ξεχωριστή συνάντηση για το θέμα αυτό όταν θα έχω κάποιες ενημερώσεις και θα εγκριθεί η επόμενη έκθεση και κάποιες ε, βεβαίως ε, κάποια νεότερα. Λοιπόν, ξέρετε, μια που έχετε ασχοληθεί και εσείς με το θέμα της αμοιβαιότητας της ΒΙΖΑ ότι ε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Εργαζόμαστε επί του ζητήματος, δίνουμε τις πιέσεις για να βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα τα πέντε κράτη-μέλη να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσει. Παραδείγματος χάρη, αυτές που αφορούν την ε, συνεργασία στον τομέα της ασφαλείας για να μειωθεί ο αριθμός απορρίψεων όπως αυτό αναφέρεται άλλωστε στην Αμερικανική νομοθεσία. Εργαζόμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία με στόχο τα αποτελέσματα. Οι ΙΠΑ επίσης είναι προσιλωμένες στο να δεχτούν τα πέντε κράτη-μέλη στο πρόγραμμα όταν μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που ορίζει η Αμερικανική νομοθεσία οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το πολιτικό κλίμα που προσανατολίζεται στην ασφάλεια στην Ουάσιγκτον δεν είναι το πιο ευνοϊκό για, για να έχουμε μια βραχυπρόθεσμη πρόοδο. Όμως, όπως είπα, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για πλήρη αμοιβαιότητα. Ο μηχανισμός αμοιβαιότητας απαιτεί η Κομισιόν να λάβει υπόψη τις συνέπειες ε, της διακοπής αυτής για τις εξωτερικές μας σχέσεις. Εμείς βεβαίως σεβόμαστε την νομοθεσία, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια ευθύνη να λάβουμε υπόψη τις αρνητικές συνέπειες. Η θέση μας παραμένει ότι δεν θα διστάσουμε να εγκρίνουμε μια πράξη κάτω εξουσιοδότηση αν αυτό βεβαίω θα οδηγήσει σε κάποια πρόοδο. Όμως, το να την ε, εγκρίνουμε αυτή τη στιγμή θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα που είχαμε επιτύχει με τον Καναδά και άλλους δείχνουν ότι η αυτή πρόοδος προς την πλήρη αμοιβαιότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεχών επαφών και βεβαίω ε, διπλωματικής εργασίας. Σκοπεύουμε λοιπόν να έχουμε μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει σε αποτελέσματα για τα 5-7 κράτη-μέλη. Όπως είπα, συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Ας το συζητήσουμε λοιπόν στην επόμενη έκθεση μας. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ε, ενισχυμένης ε, πλειοψηφίας για το πακέτο του ασύλου. Ε, διάβασα την επιστολή που αποστήλατε στον πρόεδρο Γιόνκερ. Φρανκ, Κλοντ, ήδη εδώ και τέσσερις μήνες εγώ ζητάω να υπάρξει μια συμφωνία για το θέμα το γνωρίζετε. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σημειωθεί πρόοδος γρήγορα. Έχουμε τα Συμβούλια δικαιοσύνη και Εσωτερικών αργότερα αυτή την εβδομάδα στο Λουξεμβούργο και είμαι αισιόδοξο ότι θα σημειωθεί πρόοδος εν ώψη και της συνάντησης των ηγετών την επόμενη εβδομάδα. Η Αυστριακή Προεδρία κάνει επίσης ό,τι μπορεί Τώρα, για το θέμα της μπλε κάρτας. Με την κατάλληλη πολιτική βούληση θεωρώ ότι μπορούμε να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Έχουμε έναν πολύ έμπειρο εισηγητή, τον Κλοντ, και εξαιρετικούς γεωδησηγητές. Πώ μπορούμε να αποτύχουμε. Καλούμε ιδιαίτερα στο Συμβούλιο να επανεξετάσει την θέση του έτσι ώστε η μπλε κάρτα να γίνει ένα ελκυστικό πανευρωπαϊκό σύστημα που θα προσελκύει τους ε, κατηρτισμένους εργαζόμενους που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των οικονομιών μας. Μάλιστα, η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ελλείψεων που αντιμετωπίζουμε σε κάποια επαγγέλματα σημαίνει ότι μια συμφωνία απαιτείται. Η πρότασή μας περιέχει αρκετή ευελιξία για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να την προσαρμόσουν στην αγορά εργασίας τους, δημιουργώντας ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό σύστημα για τους ειδικευμένους εργαζόμενους. Οπωσδήποτε τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να αποφασίσουν πόσους υψηλά διδικημένους εργαζόμενους χρειάζονται. Θα θέσω αυτό το ζήτημα και την Παρασκευή στο Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερικών. Κυρία Τσίπελ, θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχω ήδη πει δημοσίω και εδώ δεν είμαστε υπέρ της επαναφοράς των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων, γιατί αυτό είναι ένα βήμα προς τα πίσω για την Ευρώπη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα εν λόγω κράτη-μέλη για να καταργηθούν σταδιακά οι εσωτερικοί έλεγχοι και να αντικατασταθούν με άλλα μέτρα, όπως αστυνομική έλεγχη και διασυνοριακή συνεργασία. Όπως ήδη είχαμε προτείνει τον Οκτώβριο του 2017. Είμαστε σε στενή επαφή με τις έξι χώρες Σέγγεν που αυτή τη στιγμή διεξάγουν προσωρινούς ελέγχους. Ο στόχος μας είναι και παραμένει ο ίδιος να επανέλθουμε σε μια περιοχή Σέγγεν που θα λειτουργεί πλήρως το συντομότερο δυνατόν. Και τόνισα πριν, η προτινόμενη πρότασή μας δεν έχει στόχο να νομοποιήσει τις υφιστάμενες πρακτικές. Η πρότασή μας περιείχε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Δηλαδή, μεγαλύτερα χρονικά όρια για να ανταποκριθούμε στις θεμητές ανησυχίες των κρατών μελών που επηρεάζονται περισσότερο από τις απειλές η εισαγωγή προσωρινών εσωτερικών ελέγχων όμως πρέπει να παραμείνει ένα εξαιρετικό μέσο, μια τελευταία λύση. Ο αντίκτυπος στην ελεύθερη μετακίνηση θα πρέπει να είναι περιορισμένος και θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικά μέσα κατά προτεραιότητα όπως η αστυνομική έλεγχη. Επιπλέον δικλείδες ασφαλείας είναι ότι τα κράτη-μέλη θα αξιολογούν τακτικά τους ελέγχους αυτούς και θα συνεργάζονται με άλλα κράτη-μέλη και δεν θα προχωρούν σε μέτρα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Για το θέμα το οποίο είπατε για την ανάγκη 10.000 συνοριοφυλάκων. Οι προτινόμενοι 10.000 Ευρωπαίοι συνοριοφυλακές θα βασιστούν ήδη στον μηχανισμό που υπάρχει και το ενδεικτικό επίπεδο δεσμεύσεων των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τα άτομα τα οποία προβλέπονται στον μηχανισμό είναι πάνω από 7.000. Οι ικανότητες αυτές συμπληρώνονται από 1.500 συνοριοφύλακες που έχουν υποβάλει σε αυτήν την δεξαμενή προσωπικού τα κράτη-μέλη και οι ανάγκες σε αυτόν τον τομέα αυξάνονται. Η υπηρεσία θα χρειαστεί μόνο να στηρίξει περαιτέρω τα κράτη-μέλη αλλά να ε, κάνει επιχειρήσεις και σε τρίτες χώρες και να ενδύνει τον ρόλο της στις επιστροφές. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτό. Τώρα η κατάσταση στην ε, Μόρια. Ε, έχω έναν επιπλέον λόγο να είμαι ευαίσθητος για το θέμα αυτό. Κατ' επανάληψη είχαμε ειδοποιήσει τις ελληνικές αρχές για την κατάσταση στη Μόρια και είχαμε πει ότι είναι επίγον να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Πάντα βεβαίως είχαμε φροντίσει να υπάρχουν και διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Είμαστε σε στενή επαφή με τι ελληνικέ αρχέ για να συζητήσουμε τον καλύτερο τρόπο για να διορθωθεί η κατάσταση και να βελτιωθούν οι συνθήκε. Είχα ξαναπάει στην Ελλάδα πριν από 15 μέρε για να συζητήσω τα θέματα αυτά με τι ελληνικέ αρχέ, Συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό και όλου του αρμόδιους υπουργού. και επιτέλους καταλήξαμε σε μια συμφωνία ότι πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αλλάξει η κατάσταση γιατί όπως έχει αυτή τη στιγμή είναι ντροπή για όλους μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές ορίζοντας ότι η γενική ευθύνη για την διαχείριση των ροών στην Ελλάδα και στα hotspot ε, ανήκει βεβαίως στο ελληνικό κράτος. Ε, μιλώντας για τα hotspot, για τα όσα είπε η κυρία Σπινέλη, για τα αν τα χρειαζόμαστε ή όχι. Ε, φαντάζεστε τι θα είχε συμβεί αν δεν τα είχαμε αν ε, τα hot spot ε, υπήρχαν στην αρχή της ε, κρίσης θα είχαν πολύ καλύτερη διαχείριση. Τα, διαβάζω συχνά Η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο hot spot, η Ιταλία ένα μεγάλο hot spot. Δεν ξέρουν τι είναι. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές τι είναι. Χρειάζονται όλες αυτές οι υπηρεσίες. Eurodac, Europol, Eurojust να βρίσκονται εκεί τόπου και να κάνουν μια αξιολόγηση της κατάστασης. Είναι καλύτερο που υπάρχουν λοιπόν και μπορώ να σου πω ότι υπάρχει καλύτερη διαχείριση της κατάστασης γιατί τα hot spot έχουν αποτέλεσμα 95% των ατόμων που περνάνε το Αιγαίο δακτυλοσκοπούνται και καταγράφονται. Το ίδιο και στην Ιταλία. Ναι, ναι. Θα, θα με σταματήσετε, ο πρόεδρος. Όχι, ε, για και τα λοιπά μπορούμε να, να μιλάμε ώρες. Γιατί πολλοί από εμά έχουμε πάει εκεί, οπότε δεν θέλω τώρα να σας ε, ταλαιπωρήσω γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Θα επανέλθω αργότερα λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Λοιπόν, συνάδελφοι, ας δούμε το τι συμβαίνει εδώ. Έχουμε τόσα τεράστια θέματα και δεν είναι ικανοποιητική συζήτηση βεβαίω και για τι δύο πλευρέ γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Οπότε ας δούμε τα βασικά. Κατόπιν λοιπόν ο κύριος Κολλιό, δύο λεπτά σας παρακαλώ ο καθένας. Κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο σύντομε παρατηρήσει. Πρώτον, να καλωσορίσω τι ενέργειε ε, του Επιτρόπου και ε, να σας επενέσω για την περάσπιση του Παγκοσμίου Συμφώνου που υπερασπιστήκατε σε ολόκληρο τον κόσμο και εκεί είναι περιορισμένες οι δυνατότητές σας γιατί πολλέ ε, πολλές χώρες είναι κατά μια τέτοια ε, συμφωνία. Ε, τώρα, δεύτερα, όσον αφορά τον επίγοντα χαρακτήρα, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η πρόθεση της Κομισιόν. Υπάρχει μια προσωρινή συμφωνία επιτάπητος για το νέο, τη νέα υπηρεσία, το νέο οργανισμό για το άσυλο από τον περασμένο Ιούνιο. Δεν ε, αντιδράουμε απλά μόνο και μόνο λόγω του Συμβουλίου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τι περιμένουμε για την έγκριση του κανονισμού και έπειτα για τις υπηρεσίες, τα συστήματα μάλλον πληροφοριών. Μόνο το σύστημα Σέγγεν αποδίδει έγκαιρα και ανταποκρίνεται στις ανάγκε των πολιτών. Εγώ τώρα ως εισηγητής για το ΦΙΣ μπορώ, προσπαθώ να κάνω το ίδιο, να, δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σύστημα το οποίο να είναι πιο αποδοτικό και να ανταποκρίνεται στους στόχους του. Σήμερα είδα ε, στις εφημερίδες ότι η Κομισιόν ζητά εντολή μέχρι το τέλος του χρόνου. Εμένα με κάνει αυτό να αναρωτιέμαι. Προσπαθεί για καλύτερο χώρο έγκαιν για τους πολίτες η Κομισιόν ή προσπαθεί απλά να εξασφαλίσει το κληροδότημά της είμαστε σαφείς ότι το σύστημα αυτό δεν είναι αυτός σκοπός. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα εγκρίνουμε ένα καλύτερο σύστημα που θα βελτιώσει τη λειτουργία του Σέγγεν, θα εγγυάται καλύτερα τα δικαιώματα των πολιτών, των υπηκών των χωρών και θα αυξήσει και την ασφάλεια των πολιτών. Είστε στον ίδιο δρόμο. Ευχαριστώ για τη συντομία σας κύριε Κοέλιο. Όχι πάνω από δύο λεπτά παρακαλώ όλοι. Κυρία Σας ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε, Επίτροπε. Θα πρέπει να πω ότι δεν ε, τα βρήκατε εύκολα μπροστά σας στη διάρκεια της θητείας σας, ιδιαίτερα όσον αφορά τι μεταναστευτικές ροές. Ο αριθμός των μεταναστών που εισήλθε στην Ένωση ε, σύμφωνα με πρόσφατες, ε, πρόσφατη ενημέρωση αυξάνεται και πάλι και αυτό λόγω πιέσεων από πλευράς της Τουρκίας. Δίνουμε άπειρα χρήματα στην Τουρκία για να περιορίσει τις ροές και για να τιμωρήσει τους διακινητές. Όμως οι διακινητές βρήκαν άλλους δρόμους, Λιβύη, Λιβύη Ιταλία και βλέπουμε επίσης και τη δουλειά που γίνεται στη Λιβύη για να βοηθηθούν οι συνοριοφύλακες, οι ακτοφυλακοί για να εμποδίσουν τους διακινητές πάνω κάτω λειτουργεί. Όμως βλέπουμε και μεγάλο αριθμό μεταναστών που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική προς την Ισπανία. Και εντωμεταξύ η Ιταλική κυβέρνηση αντιδρά και ε, κύριε Βραμόπουλε, εμείς τι θα κάνουμε, περιμένουμε μεταρρύθμιση του κανονισμού του, για, του Δουβλίνου, η ευρωπαϊκή πρόταση για υποχρεωτικές και δεσμευτικές ποσοστώσεις ε, για τα κράτη-μέλη για να δεχτούν ε, τους πρόσφυγες, τι περιμένουμε να γίνει από μόνη της ως διαμαγείας. Έχουμε ακόμα περισσότερους μετανάστες, ακόμα περισσότερους πρόσφυγες. Πρέπει να σταματήσουν να περνάνε την Μεσόγειο όπου πολλοί χάνουν τη ζωή τους. Α σκεφτούμε και τι έκανε η Αυστραλία, να βρούμε μια λύση. Δηλαδή μπορούν οι μετανάστες να ζητούν το άσυλο σε μια τρίτη χώρα δηλαδή κέντρα υποδοχής τα οποία εγκαθίστανται σε τρίτες χώρες και αν το κάνουμε αυτό θα μπορέσουμε να εμποδίσουμε τους διακινητές να κερδίζουν ε, χρήματα και θα σταματήσουμε τις ροές ε, λαθρέων μεταναστών και θα μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο Πίτερ Νίτερμιλλερ. Παρακαλώ δύο λεπτά έκαστος. Σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, που είστε σήμερα μαζί μας. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι το να συζητάμε για ένα νέο σύστημα ασύλου δεν είναι πρόβλημα το οποίο ε, μας απασχολεί μόνο εμάς, αλλά κυρίως είναι το πρόβλημα που μπλοκάρει στο Συμβούλιο γιατί κάποια κρατημέλη δεν έχουν σκοπό να βρουν κοινή ευρωπαϊκή λύση και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί ε, στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο διαγράφονται ξεκάθαρη στρατηγική και την περιγράφεται πολύ καλά και στη δική σας ομιλία. Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή. Το, από την άλλη πλευρά πρέπει να πω, όλοι γνωρίζουμε πως... Ε, υπάρχει αυξανόμενη, ε, αυξανόμενη πολιτική χειραγώγηση των αριθμών των μεταναστών, της μεταναστευτικής πολιτικής, γενικά του θέματος ε, των προσφύγων. Είναι όμως πολύ κρίσιμο το θέμα και πραγματικά πολύ θα ήθελα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν όμως άλλα δύο θέματα που πρέπει να αναφέρω οπωσδήποτε. Ε, μιλήσαμε για πολύ για διαχείριση συνόρων, αλλά σχεδόν ποτέ δεν μιλάμε για τη σημασία της κοινωνικής ένταξης. Και η κοινωνική ένταξη είναι θέμα των κρατών μελών, το ξέρω. Από την άλλη πλευρά όμως χρειάζεται και ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο για την κοινωνική ένταξη και πολύ περισσότερη οικονομική στήριξη για την κοινωνική ένταξη από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Και βέβαια και πάλι και επιστροφή είναι σημαντική. Κατανοώ τι πολιτικέ συνέπειε αυτών, αλλά όταν μιλάμε για επιστροφέ θα πρέπει να μιλήσουμε και για επανένταξη όλων αυτών των ανθρώπων στην χώρα τους, στην πατρίδα τους. Γιατί κάποιες φορές ζουν δύο-τρία χρόνια εκτός της χώρας τους και πρέπει να στηρίξουμε τον κόσμο αυτό και στην επανένταξή του. Ευχαριστώ Πίτερ, Σιλβί Γκυγιώμα. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θέλω να σας πω εξ αρχής ότι συμμερίζομαι απόλυτα τα όσα είπε ο, συν, ο Πρόεδρος ε, ε, Κλόντ Μωράης για την ε, υπομονή του Ευρωκοινοβουλίου. Εσείς με μεγάλο ενθουσιασμό μιλάτε, όμως φαίνεται πως οι συνάδελφοι του Συμβουλίου δεν έχουν πρόθεση να προχωρήσουν. Έχουμε κάνει ένα σωρό εκθέσεις για να συζητήσουμε ε, το τι θα πρέπει να, και επαφέ ε, μετά από το Συμβούλιο Κορυφής του Ιουνίου. Ωστόσο είναι στήρες γιατί κυρίως ε, οι αποκλήσει διαφάνηκαν σε εκείνη τη διάσκεψη κορυφής. Έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση με την μεταναστευτική αλλά και κυρίως πολιτική κρίση. Εσείς που συμμετέχετε στις επαφές της Λιών που είναι και η πόλη μου παρεμπιπτόντος. Εσείς συναντήσατε τους Υπουργούς Εσωτερικών ε, και μάλιστα ε, έλειπε και ο Υπουργός Εξωτερικών που δεν έχει αντικατασταθεί μέχρι και σήμερα. Ε, εσείς τι πιστεύετε για την κοινή δράση ανάμεσα στη Γαλλία και την Αλία στην Ιγυρία. Θα βοηθήσει αυτό στο να αυληθούν οι βαθιές αποκλήσεις που έχουν αυτές οι δύο χώρες στην υποδοχή των ε, μεταναστών. Τι αξιόπιστο περιμένετε με τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου και ποια είναι η θέση σας για την παρουσία ανθρωπιστικών σκαφών στην Μετεσόγειο και την παρεμπόδιση του σου, γιατί ε, τον ακινητοποίηση μάλλον επειδή δεν έχει πια σημαία. Please. Ευχαριστώ Σελβίο. Κύριος ε, Κώστερ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε. Εγώ θέλω να εστιάσω στην ανθρώπινη καταστροφή στην Μεσόγειο, που είναι το πιο θανατηφόρο σύνορο στον κόσμο το ποσοστό θανάτων στη Μεσόγειο είναι υψηλότερο από ό,τι ποτέ. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι το κλείσιμο των ε, λιμανιών από την Ιταλική κυβέρνηση. Ο Υπουργός Ιστορικών Σαλβίνη απαγορεύει όχι μόνο ιδιωτικά ε, σκάφη διάσωσης, αλλά ακόμα και ε, εμπορικά πλοία, φορτηγά που μπορεί να φέρουν πρόσφυγες. Ε, απαγορεύει λοιπόν να πιάσουν αυτά τα πλοία στα λιμάνια της Ιταλίας. Από τότε λοιπόν που ο Σαλβίνη ως Υπουργός Ιστορικών της Ιταλίας το ποσοστό των θανα... το... Οι θάνατοι αυξήθηκαν από 3 σε 8 ημερησίως και ο αριθμός των μη αναφερόμενων περιστατικών είναι πολύ ψηλότερο. Τι κάνει η Κομισιόν ώστε να εξασφαλίσει ότι η Ιταλική κυβέρνηση θα κάνει το καθήκον της και θα ανοίξει πάλι τα λιμάνια της. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή τρία σωστικά ε, σκάφη, τα οποία διευθύνουν ε, ΜΚΟ, έχουν συλληφθεί στη Μάλτα και κινητοποιηθεί χωρίς νομιτική βάση. Εγώ πήγα εκεί την περασμένη εβδομάδα. Οι θελοντές αυτοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να σώσουν ε, πρόσφυγες που πνίγονται λίγα χιλιόμετρα πιο έξω στη Μεσόγειο. Κύριε Βραμόπουλε, τι κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι αυτά τα σκάφη θα επιστρέψουν στην ζώνη έρευνας και διάσωσης όπου, όπου πρέπει ε, να δουλέψουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Εσείς έχετε επαφές με τις αρχές της Μάλτας να δείτε με ποιες νομικές βάσεις κρατούνται και έχουν ακινητοποιηθεί αυτά τα, τα, σκάφη, το sea 3. έχουν θεωρηθεί εγκληματικά αυτά τα σκάφη, εγκληματίες αυτοί που τα λειτουργούν. Εσείς όμως είπατε και βάλατε ως υποψήφιο το, μια τέτοια οργάνωση για το βραβείο Ζαχάροφ. Τι θα κάνετε για αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρυσόγονος. Το μικρόφωνο του μιλτή δεν λειτουργεί. Α, τώρα εντάξει. Μεγάλα ποσά για την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών στις διάφορες δομές φιλοξενίας ε, και η διαχείριση των ποσών αυτών γίνεται κατά βάση από τις εθνικές κυβερνήσεις ή από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ωστόσο, η κατάσταση στις δομές φιλοξενίας φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Εσείς μόλις μας μιλήσατε για τη δομή της Μόριας, ε, την οποία τη χαρακτηρίσατε απογοητευτική. Ε, διατυπώνονται κατά καιρού κατηγορίες, μάλιστα δημόσια, για κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μήπως θα ήταν καλύτερα αν αντί να ε, αναθέτουμε τη διαχείριση στους φορείς αυτούς Αναλάμβαναν φορείς και υπηρεσίες της ίδιας της Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου ή η Κομισιόν με τις υπηρεσίες της, την αντιμετώπιση της κατάστασης στις δομές φιλοξενίας, ούτως ώστε να υπάρχει και πολύ αμεσότερος έλεγχος των ευρωπαϊκών οργάνων πάνω στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση αυτών των χρημάτων. Κύριε Πρόεδρε, ε, τρία θέματα θα ήθελα να θέσω. Κύριε Επιτροπέ, μιλήσατε για την επιστροφή παρατύπων μεταναστών. Μπορείτε να μας δώσετε έναν αριθμό πώς τέτοιοι υπάρχουν στην Ευρώπη κατά την αποψή σας και τι θεωρείτε, ε, πώς θεωρείτε θα έχουν επιστρέψει μέχρι το τέλος της ε, θητείας σας βεβαίως αυτό είναι η κασία αλλά δεύτερον πραγματικά μια απορρίσα που αναφέρατε ξανά το θέμα της μπλε κάρτας για να προσελκύσουμε ε, υψηλά ειδικευμένα άτομα. Δηλαδή θέλετε να ασκήσετε μια πολιτική ανθρωπίνων πόρων ε, που θέλετε να τους πάρετε από τις χώρες οι οποίες ε, χρειάζονται βοήθεια και τελικά να μην μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια προοπτική στον τόπο τους γιατί οπωσδήποτε χρειάζονται οπωσδήποτε σε αυτές τις ε, χώρες, πολύ περισσότερο από στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, ε, σήμερα αναφέρθηκε επίσης και το θέμα των μεταναστών στην ε, Τουρκία. Την άνοιξε εγώ είχα πάει στο Χαλέπι και συνάντησα και τον Δήμαρχο και τον διοικητή εκεί της πόλης, οι οποίοι μου είπαν ότι μέχρι το 2017 είχαν επιστρέψει 700.000 άτομα από την Τουρκία και τώρα πρέπει να είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ήδη. Οπότε τα στρατόπεδα στην Τουρκία για τα οποία μιλούσαμε για 3 εκατομμύρια άτομα οπωσδήποτε έχουν τώρα πολύ μικρότερους ανθρώπους και μήπως αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να περικοπεί τουλάχιστον κατά το 1 τρίτο και η οικονομική βοήθεια προς την Τουρκία για το σκοπό αυτό. Ο κ. Λόπης Αγγιλάρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε για αυτόν τον διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή μας. Ακούσατε από τους συντονιστές οι οποίοι μας εκπροσωπούν όλες τις πολιτικές ομάδες Για να είμαι κι εγώ λοιπόν λίγο χρήσιμο από το εξή. Είπατε ότι ο χρόνος ε, τελειώνει και πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της θητείας. Ναι, το νιώθουμε. Εμείς είμαστε υποψήφιοι στις εκλογές. Εμείς αντιμετωπίζουμε τους ε, ψηφοφόρου και θέλουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα εντός αυτής της ε, θητείας. Κάτι το θετικό. Και θα σας ζητούσα να έχετε κατά νου σε όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάσατε ότι όλα αυτά σχετίζονται το ένα με το άλλο και όλοι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Οπότε σας ζητώ να κάνετε ό,τι μπορείτε για να βρείτε μια σωστή ισορροπία γιατί υπάρχουν κάποια θέματα που αφορούν την ασφάλεια, άλλα αφορούν τη μετανάστευση, άλλα αφορούν το άσυλο. Πρέπει λοιπόν να κάνετε ό,τι μπορείτε, ειδικά στους τριμερείς διαλόγους, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό αυτό Κοινοβουλίο να έχει κάποια αποτελέσματα. Εγώ είμαι και εισηγητής, ίσως ξέρετε, στον κώδικα της Βίζας ε, και την έκθεση για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις ε, την προστασία του μεταναστών. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κάντε ό,τι μπορείτε στον τριμερή διάλογο για να έχουμε να βρούμε την σωστή ισορροπία. Αν το κάνετε αυτό, νομίζω ότι ε, όλοι θα συνεργαστούμε έτσι ώστε η εντολή αυτή και η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρουσιάσουμε στους ψηφοφόρους, τους οποίους εμείς βεβαίως αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ, Σόφι Νετφέλντ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη να πω ότι συμφωνώ πλήρως με τις ε, προσπάθειές σας για τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Αυτά από επένους Τώρα, για την αμοιβαιότητα της βίζας είπατε ότι ξέρω τι λέει ο νόμος, αλλά δεν θα τον εφαρμόσουμε γιατί έχει αρνητικές συνέπειες. Ε, θα το έχω κατά νου αυτό την επόμενη φορά που θα παραβιάσω τον νόμο. Λοιπόν, μετά, όταν μιλάμε για την βιασύνη του να περάσουμε ε, νομοθεσία. Ναι, αυτό δεν έχει σχέση με το τέλος της ε, θητείας. Μας πίεσαν να ψηφίσουμε την διατήρηση των δεδομένων, το PNR και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάθε φορά προκύπτει λοιπόν ότι η νομοθεσία αυτή δεν στέκει και δεύτερον ότι τα κράτη-μέλη δεν την εφαρμόζουν γιατί δεν υπάρχει τελικά εφαρμογή του πινάρ. Γιατί λοιπόν να πιστέψουμε τώρα την Κομισιόν όταν μας λέει ότι βιαζόμαστε. Μπορούμε να βιαστούμε λίγο περισσότερο με την εφαρμογή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που έχει καθυστερήσει και δεν ε, απασχολεί τα κράτη-μέλη. Μήπως ε, να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το μηχανισμό του κράτους δικαίου που ψηφίσαμε πριν από δύο χρόνια και η Κομισιόν δεν έχει κάνει τίποτα ακόμα. Θα μπορούσα να ε, πω και άλλα παραδείγματα. Όλα αυτά σχετίζονται. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν και καμία βιασύνη να εγκρίνουν το πακέτο ασύλου γιατί ξέρουν ότι εμείς θα εγκρίνουμε ό,τι θέλουν ε, ενώ ό,τι θέλουμε εμείς δεν θα το εγκρίνουν. Είμαστε ηλίθιοι και πραγματικά χωρίς ε, ανάστημα. Για την Σέγγεν τέλος συμφωνώ με αρκετές πατήσεις που έγιναν, αλλά έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Η Μίλα Κοσλόφσκα από την Ουκρανία είναι παντρεμένη με Πολωνό πολίτη και δεν μπόρεσε να μπει στην ζώνη Σέγγεν με ακούτε. Ναι, αλλά κάνω ερώτηση τώρα. Να τελειώσω την ερώτησή μου. Ωραία. Δεν της επετράπει να μπει στην ε, ζώνη Σέγγεν. Τώρα ε, μάλιστα η πολωνική κυβέρνηση είπε ναι την βάλαμε στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν γιατί αυτή και ο σύζυγός της ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Η Κομισιόν αρνείται να ερευνήσει γιατί λέει «Α, εμείς κοιτάμε μόνο το σύστημα». Ε, δηλαδή τι μπορεί να κάνει ο μεμονωμένος πολίτης, να πάει στο Λουξεμβούργο να τραβιέται πέντε χρόνια στο δικαστήριο. Εσείς υποτίθετε ότι προστατεύετε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Τερέζα θέλετε να μιλήσετε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, για ένα λεπτό γρήγορα. Όλοι μίλησαν περισσότερο, εγώ μόνο ένα λεπτό, τέλος πάντων. Ευχαριστώ, Επιτροπή. Να σας μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Ήθελα να σας πω το εξής. Στην δική μου περιφέρεια, μόνο Δευτέρα, Σάββατο και Κυριακή, τρεις μέρες, μπήκαν 2.000 μετανάστες. Και εγώ είμαι συνεχώς παρούσα εκεί, στην Αλχεθήρας, ε, μπαίνουν από την θάλασσα του Αλμποράν, από το στενό του Ιβλαρτάρ, ε, τραγωδίες, ε, πάρα πολύ ανήλικοι ασυνόδευτοι, δεν υπάρχουν δομές, ούτε οι νόμοι μας δεν είναι προσαρμοσμένοι σε αυτή την κατάσταση. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στην Ιταλία, στην Κατάνη και εκεί έχουν μειωθεί οι εισοδοί κατά 87% όμως στην Ισπανία, στις, στην Ανταλουσία φτάνουν 50% περισσότεροι από ό,τι πριν. Οπότε ποια είναι η άποψή σας και θα ήθελα να σας ζητήσω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει περιφερειοποίηση της χρηματοδότησης των κονδυλίων έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς να λάβουμε χρηματοδότηση κατευθείαν η Δήμη μας και η Περιφέρεια, η ανεξάρτητη περιοχή της ε, Ανταλουσίας. Ευχαριστώ. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας, αλλά ζήτησα από τον Επιτροπό και την ομάδα του αν μπορούν ε, να, περιμένουν λιγάκι, να μείνουν. Ε, πάρτε όσο χρόνο χρειάζεστε κύριε Επίτροπε. Δεν μπορώ να σας ζητήσω 10 ερωτήσεις να τις απαντήσετε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κλοντ. Θα ξεκινήσω και από εκεί που με σταμάτησες πριν. Δεν θέλω να αφήσω κενά. Σε ό,τι αφορά την συνεργασία μας με τρίτες χώρες, βασίζεται σε πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης. Έχω συναντήσει και την ηγεσία της χώρας και τους αρμόδιους υπουργούς πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ θερμό κλίμα σχέσεις μας. Χθες στη Λιόν ξανασυνάντησα τον Υπουργό Εσωτερικών του Μαρόκο και σύντομα θα ξαναεπισκεφθώ τη χώρα. Θα σας πω ότι πριν από τρία χρόνια το κλίμα των σχέσεων με τρίτες χώρες ήταν πολύ χειρότερο. Έχει βελτιωθεί και όλο και περισσότερες χώρες της περιοχής μας επιθυμούν να συνεργαστούν και συνεργάζονται. Για παράδειγμα Νιγηρία και άλλες χώρες. Εγώ επίσης να σας πω ότι ποτέ δεν επέκρινα το κοινοβούλιο, αντιθέτως. Και το κάνω σκοπό επίμως επενώ το Κοινοβούλιο γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έκανα το ίδιο κυρία Ζήπλ με το Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο, ε, το Συμβούλιο το έχω επικρίνει και πολλές φορές αυστηρά, ιδιαίτερα συγκεκριμένε κυβερνήσεις. Γνωρίζετε ε, ότι από την αρχή το βασικό μας πρόβλημα σε σχέση με τη μετανάστευση ήταν στο Συμβούλιο και το πρόβλημα αυτό έχει επιδεινωθεί. Όμως, η Κομισιόν παίζει τον ηγετικό της ρόλο. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν από τρία χρόνια, χάρη στη συνεργασία μας. Σε ό,τι αφορά τους τριμμένους διαλόγους για το πακέτο του ασύλου, η Κομισιόν σας στήριξε. Το γνωρίζετε. Αλλά όπως και εσείς και εγώ λύσεις θέλουμε. Όχι παράπονα και με ψημυρία. Ε, ζήτησα από την Αυστριακή Προεδρία να περιορίσει τις αλλαγές που θα επιφέρει και να βρει ένα συμβασμό. Μέχρι τώρα η, εργασία, η συνεργασία μας είναι πολύ επικοδομητική. Στις ε, προσπάθειες ε, ε, επανεγκατάστασης των κρατών μέλων, πρέπει να σας πω ότι από 8.000 το 2015 πέρασαμε στις 24.000 το 2017, δηλαδή τεπλασιάστηκαν τα κράτη-μέλη σε αυτήν την περίπτωση ανταποκρίθηκαν γρήγορα στη σύσταση της Κομισιόν του Σεπτεμβρίου 2015 για επιπρόσθετες 15.000 θέσεις μέχρι τον Οκτώβριο 2019 για επανεγκατάσταση. Πράγματι, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου είχαν ήδη υποσχεθεί περισσότερα από όσα είχαμε ζητήσει. Κλοντ, για το θέμα της ε, κυρίας Μπιόρκ και μετά τις ανταλλαγές μας. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε μια ανεξάρτητη πρόταση και είναι απολύτως απαραίτητο να μην χαθούν τα εφιστάμενα κονδύλια. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και θα πρέπει μια ακόμα φορά να ζητήσω από το Κοινοβουλίο να βιαστεί και να υιοθετήσει την απόφαση του μέχρι το τέλος του χρόνου. Μου η κυρία Μπιόρκ γνωρίζει ότι είμαστε έτοιμοι, ότι βασίζουμε σε αυτήν. Κάλώ για, για, το, για το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Γνωρίζω ότι οι πολωνικέ και αυστριακέ αρχέ έχουν κάνει συγκεκριμένα σχόλια. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Θα του συναντήσω στο Συμβούλιο Τζάι αργότερα αυτή τη βδομάδα και θα μιλήσω μαζί τους. Αλλά το είπα και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα. Και το ξαναλέω εδώ. Η θέση της Κομισιόν είναι σαφής. Η μετανάστευση είναι ένα, μια παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί παγκόσμιες λύσεις και παγκόσμια ε, κατανομή των ευθυνών. Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία ασύλου. Δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε άλλο. Θέλουμε να εξασφαλιστεί ότι η υπηρεσία θα μπορεί να στηρίζει πλήρως στα κράτη-μέλη, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Και το σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων, το VIS. Γνωρίζω ότι κάνετε ό,τι μπορείτε. Οι υπηρεσίες μου είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν να διευκρινίσετε οτιδήποτε χρειάζεται, διευκρίνηση στην πρότασή μας. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όπως κάνατε και με το SIS, το Σύστημα Πληροφοριών Σέγγεν σε ό,τι αφορά τους επιστρεφόμενους σε τρίτες χώρες. Η ιδέα έρχεται και ξανάρχεται στο τραπέζι. Εγώ είμαι πάντοτε σαφής. Δεν έχουμε συζητήσει αυτή την ιδέα με καμία τρίτη χώρα και δεν σκοπεύουμε κιόλας να το πράξουμε. Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, το, για τις επιστροφές είναι Σαφή και εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Οποιαδήποτε καινούργια διαδικασία θα πρέπει να εναρμονίζεται με τους υφιστάμενου κανόνες. Πίτερ, ανέφερε κάτι ιδιαίτερα εξόχως πολιτικό. Και η ασφάλεια και η μετανάστευση είναι θέματα τα οποία μπορούν να τύχουν διαφορετικής χρήσης. Δική μας κοινή πολιτική ευθύνη είναι να υιοθετούμε μέτρα που θα είναι αποτελεσματικά οι πολίτες θα πρέπει να βλέπουν τα αποτελέσματα της δουλειάς που κάνουμε εμείς εδώ μαζί. Ό,τι καταφέρουμε εμείς εδώ θα επηρεάσει και ενδεχομένως θα καθορίσει την πολιτική ατμόσφαιρα πρώτων επερχόμενων ε, ευρωεκλογών. Σε ό,τι φορά την ολοκλήρωση πρέπει να εντείνουμε τις κοινωνικές προσπάθειες. Όσο πιο πολύ στηρίζουμε τις ε, χώρες επιχειρησιακά και, οικονομικά, τόσο το καλύτερο. Ε, ξέρετε ότι έχουμε αυξήσει τα κονδύλια στο επόμενο πολιτεύει δημοσιονομικό πλαίσιο. Για το Aquarius χαίρομαι που βρέθηκε λύση, Πριν όμως θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν αρκούν οι ad hoc λύσεις, χρειαζόμαστε μόνιμες, βιώσιμες λύσεις η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητα να πει πού θα πρέπει να ε, την χάνουν υποδοχή στα πλοία. Όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου η Κομισιόν στις Ιουλίου ε, δημοσίευσε ένα εγγραφό για τις ε, περιφερειακές πλατφόρμες και τα κέντρα ελέγχου. Με πολύ σαφήνεια για τους στόχους. Ποιοι είναι οι στόχοι. Να εξασφαλίσουμε μια γρήγορη και ασφαλή ε, υποδοχή και καλές συνθήκες. Καθώς επίσης και τις αρχές οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη δημιουργία τέτοιων πλατφορμών. Σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, οι διεργασίες συνεχίζονται. Διεθνή οργανισμοί, ε, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η, η Πατιαρμοστία, συνεχίζουν τη δουλειά για να διευθυνιστεί καλύτερα ο, ο ορισμός της έννοιας. Τώρα θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας γιατί θέλω να μιλήσω στα ελληνικά, να απαντήσω στον κύριο Χρυσόγονο. Ε, αγαπητέ κύριε Χρυσόγονε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν κανόνες. Τα κράτη-μέλη είναι αποκλειστικά αρμόδια και υπεύθυνα για την εφαρμογή των πολιτικών που αποφασίζουμε εμείς. Αυτά είναι μια βασική αρχή που διέπει συνολικά την ε, λειτουργία ε, των σχέσεων ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη-μέλη. Και εμείς δεν μπορούμε να τα υποκαταστήσουμε. Θα παρατηρήσατε όμως ότι όπου υπήρχαν έκτακτες, ε, επίγουσες ανάγκες ε, και προβλήματα ε, απορρόφησης, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε πρακτικά με τη χρήση διαφορετικής διαθέσιμης πηγής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε επίγουσας ανάγκης. Αναφέρομαι εδώ στην απευθείας χρηματοδότηση διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τώρα για τη χρηματοδότηση στην Ελλάδα που αναφερθήκατε. Γνωρίζετε ότι από την πρώτη και όλα στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει στη διάθεση της Ελλάδος μια πολύ σημαντική οικονομική βοήθεια συμπεριλαμβανομένης και έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλουν οι ελληνικές αρχές για να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μεταναστευτικές ροές και να αντιμετωπίσουν τις ε, συνεπακόλουθες ε, προκλήσεις. Σήμερα, για παράδειγμα, σήμερα, παρήχαμε στην Ελλάδα ε, πλέον 24,1 εκατομμύρια ευρώ στον IOM, στον Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση, για να υποστηρίξουμε την διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, για να διασφαλίσουμε ότι παιδιά μετανάστες θα μεταφερθούν άμεσα σε ασφαλές περιβάλλον και θα τους παρέχεται εκπαίδευση. Συνολικά, η Ελλάδα έχει στην διάθεσή της 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την διαχείριση του μεταναστευτικού, της ανθρωπιστικής κατάστασης και των εξωτερικών συνόρων για το διάστημα από το 2014 μέχρι το 2020. Ε, and now I come back to και ε, τώρα επανέρχομαι στα αγγλικά. Για τις επιστροφές αυτή τη στιγμή, αφού με ρωτήσατε, οι επιστροφές πράγματι δεν είναι ικανοποιητικές. 36,6% των παρατύπων μεταναστών επιστρέφουν. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν είναι αποτελεσματικές οι διαδικασίες στο εθνικό επίπεδο και δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς ε, τα μέσα για να σταματήσει η εξαφάνιση τρινά των ε, μεταναστών. Και βεβαίως η έλλειψη επανε, ε, συμφωνίας και συνεργασίας στο θέμα της επανεισδοχής από τις χώρες προέλευσης. Έχω έρθει πολλέ φορέ σε επαφή με το Πακιστάν και άλλε χώρε. Μου υποσχέθηκαν πολλά πράγματα, αλλά τίποτα δεν συνέβη. Οπότε συνεχίζουμε τη συνεργασία με αυτέ τι χώρε. Δεν μπορώ να προβλέψω πόσοι ακόμα πρέπει να επιστραφούν. Πρέπει να είμαι ειλικρινή. Γιατί όλα αυτά εξαρτώνται από την εθνική εφαρμογή. Γι' αυτό προτείνουμε να μεταρρυθμίσουμε την οδηγία περί επιστροφών. Juan Fernando. όλοι μαζί είμαστε εδώ πέρα. Συμφωνώ, αντιμετωπίζουμε τους ε, ψηφοφόρους. Όλοι μας. Θέλουμε και θα υπερασπιστούμε την Ευρωπαϊκή μας Ένωση και τις αξίες μας. Οι πολιτικές μας. Ξέρετε ότι αυτό θα είναι τμήμα της κληρονομιάς που θα αφήσουμε εσείς και η Κομισιόν σε λίγους μήνες. Και θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε κάνει πολλά. Η κατάσταση δεν είναι αυτή που ήταν πριν από τρία χρόνια. Όλοι θυμόμαστε. Αλλά βεβαίω πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν. Και βεβαίως η προτεραιότητα μας τώρα είναι να οριστικοποιηθούν όλα αυτά τα θέματα. Είναι επίσης ευθύνη μας, πέρα από αυτό, να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες με γεγονότα και με αποτελέσματα. Σοφή, για το PNR, τα δεδομένα αεροπορικών υπατών. Ξέρω πόσο ευαισθητήσεις στο θέμα. Είδες μετά από τόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Θέλω να σας πω ότι στις 19 Ιουλίου φέτος η Κομισιόν αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάση κατά των κρατών μελών που είχαν αποτύχει να κοινοποιήσουν την πλήρη εφαρμογή μέχρι εκείνη την ημέρα. Η Κομισιόν επίσης θα ξεκινήσει μια αξιολόγηση πληρότητας ε, και συμμόρφωσης των εθνικών μέτρων μεταφοράς. Έχω κατά επανάληψη ζητήσει από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν γρήγορα ε, τα συμφωνηθέντα. Συμφωνώ μαζί σας ότι οι καθυστερήσεις είναι απαράδεκτες. Ο μηχανισμός PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταστεί λειτουργικός το συντομότερο δυνατόν. Αγαπητοί συνάδελφοι αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας. Να κλείσω αυτήν την συζήτηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι. Προσπάθησα να απαντήσω στις περισσότερες ερωτήσεις παρά το ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά αυτά τα ζητήματα. Και θα δεχτώ την πρόσκληση του Πρόεδρου Και μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μου αν χρειάζεστε τεχνική στήριξη του υπηρεσίε μου ή πολιτική, πολιτικό συντονισμό για να επιτύχουμε τον κοινό μα στόχο. επίση, αναμένω, όπως και τα τελευταία τέσσερα χρόνια, την στήριξή σας ε, και για να στείλουμε μηνύματα στο Συμβούλιο αλλά και για να μεταφέρουμε στο μέτωπο τη επικοινωνία στην δουλειά που κάνουμε στον Ευρωπαίο πολίτη. Γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν συνεργάζονται στενά για να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο. Και σας ευχαριστώ και πάλι για την συνεισφορά σας έτσι ώστε να μπορούμε σήμερα να πούμε ότι έχουμε κάνει πολλά αλλά και ότι απομένουν πολλά να κάνουμε για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπο. Να πω το εξή. Πράγματι, εγώ είμαι μάρτυρας σε αυτά. Υποστηρίζεται το Κοινοβούλιο και πάντα υποστηρίζεται τη θέση του Κοινοβουλίου. Το βλέπω ο ίδιος ε, και πρέπει να είμαι ειλικρινής ε, και να το πω ότι πράγματι συγκρούεστε με το Συμβουλίο. Έχουμε ασκητά μεγάλη μυρισιά διάταξη έχουν πολλά κοινά θέματα και βεβαίω πάντα είστε στην διάθεσή μα. Ζητώ συγγνώμη που συζητήσαμε τόσα πολλά θέματα σε τόσο λίγο χρόνο, ήταν σχεδόν αδύνατο. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Είναι μια στατική βασανιστήριο Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας σήμερα και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Να περάσει ο επόμενος επίτροπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. And the team, by the way. So, colleagues, my sincere apologies for the late start. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αγαπητοί συνάδελφοι, από τον εισηγητή και τους υπόλοιπους. η συζήτηση αυτή ξεκίνησε αργά και πήγε και ε, δεν διαχειρίστηκα πολύ αποτελεσματικά οπότε ξεκινάμε με 25 λεπτά καθυστέρηση μόλις έρθει λοιπόν ο Επίτροπος. So, colleagues, uh, we're starting very late, so no introductions from me. Ξεκινάμε με μεγάλη καθυστέρηση. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε. Θα μιλήσουμε για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Όλοι γνωρίζουν αυτόν τον νέο φάκελο. Έχουμε ορίσει η για αυτόν το θέμα, την κυρία Στίβενς. Είναι παρούσα, χωρίς άλλες εισηγήσεις από πλευράς μου. Και έχετε διαδικαστικό. Α, θέλετε να μιλήσετε. Εντάξει. Α, να είμαι πολύ κουρασμένος. Όχι, εντάξει, αστεία λέω. Λοιπόν, μην μου κουνάτε τις κάρτες απότομα μπροστά μου. Χωρίς άλλες ε, λοιπόν εισηγήσεις και ζητώ συγγνώμη που αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Επίτροπε, δικό μου στο λάθος, οπότε... Να ακούσουμε τη δική σας ε, εισήγηση για το νέο φάκελο για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου online. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένα σωρό επίτροποι σας ενοχλούν ε, απόψε, αλλά είναι μια σημαντική ευκαιρία να έχουμε μια πρώτη σύντομη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και ίσως να πω και δύο λόγια για μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας ε, κατά τη διάρκεια των εκλογών. Το συζητήσαμε με κάποιους από εσά σε άλλο πλαίσιο, αλλά νομίζω πως θα έχει ε, νόημα να το συζητήσουμε και ενώπιον της Επιτροπής. Θα γνωρίζετε, γιατί το έχουμε ε, συζητήσει παλιότερα, πως αυτή η πρόκληση της ριζοσπαστικοποίησης είναι ο πυρήνας της δουλειάς μας ασφάλειας, ότι δηλαδή η πρόληψη είναι πάντοτε καλύτερη από τη θεραπεία. Κάνουμε μια σειρά από πράγματα ε, για την, κατά της ριζοσπαστικοποίησης ε, offline στις κοινότητές μας και μάλιστα με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο έχουμε μια, ένα νέο γύρο ε, για το νέο ενισχυμένο κύκλο μέτρων που πρέπει να λάβουμε για να ενισχυθεί η ε, προσπάθεια αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης στις κοινότητές μας, στις ε, πόλεις μας. Ε, όμως η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα online είναι ότι άνθρωποι χωρίς να έχουν πάει στο Ιράκ, στη Συρία ή σε άλλες περιοχές σύγκρουσης, ε, μέσα στις ίδιες τους κοινότητες και στα σπίτια τους τα ίδια ριζοσπαστικοποιούνται γιατί καταναλώνουν μια τεράστια μάζα τέτοιου περιεχομένου. Κάθε μία από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια είχε μια διάσταση περιεχομένου online σε ορισμένε περιπτώσεις μέσω οδηγιών και σε πολλές περιπτώσεις λόγω της, ε, ε, του, του δοξασμού αυτής της υπέροχης κατάστασης. Και πρέπει αυτό το, να το χειριστούμε λοιπόν. Η πρόκληση είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Είναι αλήθεια ότι με την ε, πτώση των οχυρών ε, του Νταές στη Συρία, οι δυνατότητες τους για να, να φτιάξουν πολύ ε, επαγγελματικό υλικό μειώθηκε. Ωστόσο, 700 ε, ε post ε, του ΝΤΑΕΣ αναρτήθηκαν ε, παρόλα αυτά μέσα στο πρώτο εξάμεινο αυτού του έτους. Σε λιγότερο επαγγελματικό επίπεδο υπάρχουν και άλλα που αναρτώνται από ανθρώπους εδώ στην Ευρώπη, από άτομα εδώ στην Ευρώπη που εξακολουθούν να είναι ισχυρά ακόμα και αν δεν είναι τόσο επαγγελματικά και επηρεάζονται εκατοντάδες πλατφόρμες. Οπότε η Europol πρέπει να μπορέσει να αντιμετωπίσει το τρομοκρατικό περιεχόμενο σε 150 πλατφόρμες τουλάχιστον. Σε μια μελέτη του Υπουργείου Ιστορικών της Βρετανίας είδαν ότι το ΝΤΑΕΣ στηρίζει υλικό σε πάνω από 400 πλατφόρμες. Είχαμε λοιπόν ε, καλή συνεργασία στο πλαίσιο ε, του, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ιντερνετ. Εξαιρετική ιδέα και οι μεγάλες εταιρείες ε, τόσο τους άρεσε που το αντέγραψαν και έφτιαξαν το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Ιντερνετ. Ειδικά για, εκεί μπορέσαμε να δούμε με μεγάλες εταιρείες δεν μπορούν να κάνουν επιθελοντικές βάσεις και πρέπει να αναγνωρίσω ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν ε, καταβάλει προσπάθεια γιατί κατάλαβαν πόσο μεγάλος κίνδυνος υπάρχει για τη φήμη τους και κάναν διάφορα πράγματα συμπεριλαμβανομένες ε, της χρήσης κάποιων αυτοματοποιημένων μέτρων που έχουν κάτι κάνει, ωστόσο παραμένει μεγάλη προσπάθεια και μετακινείται αλλού. Αν κανείς το πετύχει στις μεγάλες πλατφόρμες μπορεί να μεταφερθεί και στις μικρότερες. Αλλά και ακόμα από τις μεγάλες πλατφόρμες αλλά και από τις μικρομεσαίες ότι έχουν να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις για την αντιμετώπιση αυτού του υλικού. Εάν είσαι μεγάλη πλατφόρμα έχεις χρήματα, μπορείς να προσλάβεις χιλιάδες κόσμου να φτιάξεις μια ομάδα που δουλεύει γι' αυτό 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείς να, να εφαρμόσεις τους όρους και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικά και να έχεις εμπιστοσύνη στην στι αποφάσει που λαμβάνει. Όταν όμω είσαι μια μικρότερη πλατφόρμα και κάποιε από αυτέ είναι αρκετά μικρέ, ε, τότε είναι πολύ πιο μεγάλη πρόκληση αυτή η υπόθεση. Και ανησυχούν ότι απλά αν εφαρμόσουν του όρου και τι προποθέσει, ακόμα και όταν ε, βοηθηθούν, ε, μένουν εκτεθειμένοι και σε νομικές δηλαδή ε, ε, διώξεις ή προκλήσεις. Και γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε την εθελοντική βάση την οποία έχουμε και την συνεχίζουμε και στο Παγκόσμιο Φόρουμ για το ίντερνετ μας, με μια, πρέπει να το ενισχύσουμε με μια νομοθεσία που να θεσπίζει μια ροή, μια βασική δηλαδή προσέγγιση νομικά ξεκάθαρη και ε, εφαρμοστέα για όλους. Και αυτό προσπαθήσαμε να προωθήσουμε με τούτη μας την πρόταση που τώρα έχετε ενώπιόν σας προσπαθεί να δημιουργήσει τρεις νέες ε, ε, υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις, ε, υποχρέωση καταρχάς στα κράτη-μέλη, ώστε να εξασφαλίσουμε πως έχουν τις απαραίτητες και προσιλωμένες δυνατότητες για την επιβολή του νόμου με παρκείς πόρους και στελέχωση για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Αρκετά κράτη-μέλη το έχουν ήδη, ειδικά εκείνα που ήδη έχουν δεχτεί επιθέσεις στους δρόμους τους που συνδέονται με ε, περιεχόμενο τρομοκρατικού χαρακτήρα ε, στο ε, διαδίκτυο. Όμως δεν, το έχουν, δεν, έχουν, δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένα όλα τα κρατημέλη και το πρόβλημα εξορισμού είναι κινητό. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος, εκεί θα πάει το υλικό. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε σαφή υποχρέωση στα κράτη-μέλη να αναλάβουν αυτή τη δουλειά. Ε, δεύτερον, ε, και αυτό είναι νέο, θέλουμε να επιβάλλουμε υποχρέωση στις ίδιες τις πλατφόρμες με ισότιμο τρόπο σε όλες τις πλατφόρμες, ώστε οι αρχές επιβολής του νόμου, οι δικαστικές, οι νομικές αρχές, όταν εντοπίζουν ένα υλικό που είναι παράνομο, σύμφωνα με σαφώς καθορισμένο ορισμό, που θα φτιάξουμε ε, και θα συμπεριλάβουμε στην νομοθεσία μας θα ε, πρέπει να κινήσουν νομική διαδικασία ε, και η, πλατφόρμα θα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει και να αφαιρέσει το εν λόγω υλικό εντός μιας ώρας. Αυτό το περιχαρακώνουμε με συγκεκριμένες στεναρές ε, δυνατότητες ε, ε, καταγγελίας ή έφεσης. Δεν φαντάζομαι βέβαια ότι οι τρομοκράτες θα χρησιμοποιήσουν το δυνατότητα καταγγελίας, αλλά είναι σίγουρο ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και πρέπει να έχουμε διατάξεις σε περίπτωση που προκύψουν κάποιες τέτοιες πιθανότητες. Οι μικρές πλατφόρμες λένε ότι αυτό θα τους βοηθήσει πολύ γιατί αφαιρείται έτσι δική τους υποχρέωση να προβούν οι ίδιοι σε κρίση με βάση τις όρους και τις ε, προϋποθέσεις τους επί των οποίων μετά θα μπορούσαν να διωχθούν. Τι κάνουν, θα επιβάλλουν μία ε, ε, νομική επιταγή που τους επιβάλλεται από τα κράτη. Και επίσης αυτό οδηγεί σε μεγάλη διαφάνεια. Τρίτη υποχρέωση που προτείνουμε είναι αν η πλατφόρμα σου, οποιοδήποτε μέγεθος και αν έχει, μπορεί αποδεδειγμένα, μάλλον χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα ώστε να μετακινηθεί περιεχόμενο τρομοκρατικό από τον ΤΑΕΣ ή κάποιον άλλο οργάνωση που βάζει λοιπόν ε, τρομοκρατικό υλικό ε, στη δική σου πλατφόρμα, τότε οι αρχές θα έρθουν σε επαφή με την πλατφόρμα και θα συμφωνήσουν για ένα σύνολο μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν ε, για να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι χρησιμοποιείται αυτή η πλατφόρμα. Αλλά αυτά θα φτιάχνονται αναπερίπτωση, δηλαδή δεν είναι μια γενική και ομοιόμορφη εφαρμογή, είναι μια αναλογική προσέγγιση ώστε να αντιμετωπίζονται τα εντοπισμένα και συγκεκριμένα προβλήματα κάθε φορά και πάλι με στεναρές ασφαλιστικές δικλίδες για δυνατότητες ε, νομικής προσφυγής. Άρα λοιπόν να τα βάλουμε όλα μαζί ε, δημιουργείται ισότιμο πεδίο, είναι το ίδιο για όλους. Δεύτερον, υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια για τα κράτη-μέλη και τις εταιρείες, διότι και οι δύο χρειάζεται να αναφέρουν τι προσπάθειες καταβάλουν και να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας. Κατά κάποιο τρόπο αυτό ε, καθησυχάζει και εξασφαλίζει περισσότερο όλους όσοι συμμετέχουν. Περιμένουμε βέβαια ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πλατφορμών θα συνεργαστούν. Αλλά πρέπει να προβλέψουμε και τη δυνατότητα κυρώσεων. Και γι' αυτό είπαμε ότι αυτές οι κυρώσεις θα πρέπει να ορίζονται ε, με συζήτηση με τα κατημέλη σε ισχυρότερη περίπτωση πλήρους και συστηματικής αποτυχίας συμμόρφωσης και θα μπορούσαν δυνατικά να ανέλθουν στο 4% του κύκλου εργασιών που κάτι το οποίο μας γνωστό από την οδηγία της GDPR. Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως μηχανισμός για να κερδίζουμε ε, χρήματα γιατί θέλουμε να ε, τις ξεγελάσουμε, να του εκμεταλλευτούμε, αλλά θα πρέπει να σκεφτείτε ένα ε, σύστημα βαθμιαίων κυρώσεων, ας πούμε, ώστε να μπορούν να ε, ε, χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το τι κάνει καθένας. Δεν πρόβλημα ότι θα έχουμε πολλές περιπτώσεις συστηματικής μη συμμόρφωσης μπορεί που και που να γίνει κάποιο λάθος, αλλά συστηματικά να μην συνεργάζονται με τις αρχές για αυτά τα θέματα οι πλατφόρμες δεν το φανταζόμαστε. Αν όμως υπάρξει τέτοια περίπτωση, αν υπάρξει μια πλατφόρμα που συστηματικά αδυνατεί ή δεν θέλει να συμμορφωθεί, θα υπάρχει δυνατότητα επιβολής ε, ε, κυρώσεων δεδομενη της απειλής. Λυπούμε που σχετικά αργά ήρθαμε με μια τέτοια πρόταση, σα υποβάλαμε αυτή την πρόταση, αλλά θέλαμε να έχουμε συγκεκριμένη, στοχοθετημένη και ε, έτσι, συγκροτημένη πρόταση και γι' αυτό θέλουμε τώρα να συνεργαστούμε μαζί σας με την συγχύτρια, την κυρία Στίβενς, τους ε, Σκιώδης, που νομίζω τώρα ορίζεται, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε γρήγορα αν μπορείτε να εικονίσετε και να εγκρίνετε την έκθεσή σας όσο γίνεται πιο σύντομα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ήδη φέτος τη συζήτηση στο Συμβούλιο για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτήν την πολύ σημαντική νομοθεσία εντός της τρέχουσας θητείας. Αν μου επιτρέπετε δύο λόγια για την ασφάλεια των εκλογών, γιατί δεν θέλω να μην το έχω αναφέρει αυτό στην Επιτροπή σας. Το τρομοκρατικό περιεχόμενο online είναι ε, ένα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, αλλά μόνο ένα ε, από τα κακά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, στο διαδίκτυο. Η χρήση μέσων επί διαδικτύου για να χειραγωγήσει κανείς τη δημοκρατική ζωή μας ή να παρέμβει στη δημοκρατική ζωή μας, στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημοκρατικές διαδικασίες είναι ε, πραγματικά κάτι πολύ ανησυχητικό και υπάρχει πολύ ε, λαϊκή ανησυχία για αυτό το θέμα, ε, δηλαδή ο κόσμος ανησυχεί, περιμένουμε ευρωεκλογέ, σε κάποιες, άλλες, σε κάποιες χώρες υπάρχουν και κοινοβουλευτικέ εκλογές και έχουμε και τις ευρωεκλογέ όπως είπαμε, οπότε Έχουμε προβεί σε κάποια βήματα ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια πτυχές του προβλήματος. Όπως ξέρετε, ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της, Ευρω... της Ένωσης ε, μίλησε για διάφορες πτυχές ε, της ασφάλειας στο διαδίκτυο ε, μέτρα για την κυβερνό ασφάλεια ενάντια σε επιθέσεις παραδοσιακού τύπου επί των συστημάτων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στις ε, διάρκεια εκλογών. Έχουμε κάνει κάποια πρόοδο με το δίκτυο νης κυβερνοεμπειρογνωμόνων που μας δέδωσαν ε, κάποιες προτάσεις τις οποίες μελετούμε Επίσης ε, χειραγώγηση, hacks, ε, διαρροές, ε, ψευδείς ειδήσει, fake news που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια άλλη σειρά θεμάτων εκεί όπως και η ανάπτυξη με, με τον Επίτροπο Γκαμπριέλ για την ανάπτυξη μεγαλύτερης διαφάνειας και λογοδοσίας το διαδίκτυο, κώδικας δεντολογίας για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, που συμφωνήσαμε διεθνώς με τις μεγαλύτερες πλατφόρμες, αυτό ήταν, ήμασταν οι πρώτοι, και έπειτα κατάχρηση προσωπικών ε, δεδομένων. Για, εκεί εστιάζουμε στο πώς ε, ε, χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα για την μικροστόχευση μέσω πολιτικού περιεχομένου. Αυτό μέσω διαπραγματεύσεων με τις πλατφόρμες που προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και έπειτα με διάφορα μέτρα με τα πολιτικά κόμματα. Περιλαμβάνονται αυτά και στη δέσμη του Προέδρου Γιούνκερ, αυτά σε συνεργασία με την Επιτροπό Γιουρόβα. Ένα σημείο που σύντομα θα πρέπει να τροποποιήσουμε είναι η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων ώστε να είμαστε βέβαιοι πως τα ευρωπαϊκά κόμματα θα έχουν και θα προστατεύουν μέτρα, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και εκείνα. Τώρα, για το Facebook και το ψήφισμα που εγκρίνατε πριν από λίγο, διαβάζοντας το γρήγορα, δεν είδα υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε αυτά που είπατε και που είπαμε. Ίσως υπάρχουν ε, τομείς όπου θα θέλατε να προχωρήσουμε περισσότερο και βεβαίως με χαρά θα συζητήσουμε μαζί σας για όλα αυτά τα θέματα. Ο Πρόεδρος, ε, κάποιοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Η κυρία Στίβενς αρχικά, ως εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλό απόγευμα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κιν και την ομάδα του για την πρόταση αυτή. Η καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας ε, σε όλες τις, τις μορφές είναι μια σοβαρή πρόκληση για όλους μας. Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στον ρόλο μου ως ε, συνεισηγήτρια έχω δει τα κενά που υπάρχουν ε, και στην νομοθεσία και στην ε, πολιτική και εξακολουθούν ακριβώς να εκμεταλλεύονται αυτά τα κενά οι τρομοκράτες. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση για όλους τους πιθανούς τρόπους διάδοσης αυτής της ιδεολογίας το Ισλαμικό κράτος, ε, η μοναδική τρομοκρατική οργάνωση ε, που έχει μια εδαφική βάση, χάνει ε, συνεχώς έδαφος από τους στρατούς στο Ιράκ και στην Συρία και έτσι αναγκάζεται να αναζητήσει άλλους τρόπους να διατηρήσει ισχύ και επιρροή και πλέον η τζιχάντ μεταφέρεται στο διαδίκτυο η διάδοση, μισους ε, οι οδηγίες ε, σε άτομα για το πώς μπορούν να σχεδιάσουν την τέλεια επίθεση είναι ανοιχτά διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Και οι πρόσφατες κυβερνοεπιχειρήσεις ε, ξεκαθάρισαν ότι δεν τα έχουμε δει όλα. Παραδείγματο χάρη στην Ολλανδία την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις αποδείξεις επίθεσης από την Ρωσία κατά του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων. Έχει φτάσει η στιγμή να κάνουμε κάτι για όλα αυτά. Μετά την φυσική ασφάλεια πρέπει να κάνουμε κάτι και για την κυβερνοασφαλή. Με μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Οπότε αναμένω όλοι μαζί να καταλήξουμε σε μια ισχυρή νομοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Χέλγα, λοιπόν, για τους ε, ήταν ε, βεβαίως ε, πολύ φρέσκο το θέμα. Η κυρία Ντατή ε, ήταν η αρμόδια. Αλλά μου έστειλε ένα σημείωμα ότι έχει κλείσει η φωνή της, οπότε θα διαβάσει τις ερωτήσεις Υπάρχει άλλη σκιώδη Η Εύα Ζολή των Πρασίνων μόλις έφυγε. Μα τι είναι αυτό το θέμα. Κάποιος άλλος σκιώδη θέλει να φύγει. Χέλγα, τι τους έκανες. Κανένας άλλος. Οπότε ξεκινάμε την κυρία Σίπελ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για την παρουσίασή του. Το τρομοκρατικό περιεχόμενο ε, δεν θα πρέπει να διαδίδεται και να επηρεάζει τη συνείδηση των ανθρώπων. Όμως ε, πολύ συχνά η πρόκληση βρίσκεται στι λεπτομέρειε. Οπότε, η ερώτησή μου, γιατί χρειαζόμαστε καινούρια πρόταση. Αν κάτι είναι ήδη παράνομο, είτε offline είτε online είτε εκτό στο ίντερνετ είτε στο ίντερνετ θα πρέπει να αφαιρείται όταν υπάρχει ένα βιβλίο που πουλιάται σε ένα βιβλιοπωλείο και έχει παράνομο περιεχόμενο θα πρέπει να αποσύρεται γιατί χρειάζεται διαφορετική πρόταση για το online περιεχόμενο δεύτερον μιλάμε για τρομοκρατικό περιεχόμενο όχι απλώς για παράνομο περιεχόμενο υπάρχει μια γραμμή διάκρισης ανάμεσα στο ένα και στο άλλο, δηλαδή στο παράνομο περιεχόμενο και στο τρομοκρατικό περιεχόμενο. Έχουμε κοινή αντίληψη για το τι σημαίνει τρομοκρατικό περιεχόμενο και το καταλαβαίνουν με τον ίδιο τρόπο όλα τα κράτη-μέλη. Μήπως υπάρχουν πράγματα που επιτρέπονται σε μια χώρα αλλά όχι σε άλλη. Μετά, λέτε ότι χρειάζεται οι αστυνομικές αρχές να έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα και γενικώ οι, οι, δυνάμεις του νόμου. Ε, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει να έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές. Μιλάτε για τεχνικές ικανότητες. Τι εννοείτε ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό που μιλάμε για ορισμούς τόσο νωρίς. Γιατί έχουμε πάρει μέρος σε πολύ λεπτομερή σεμινάρια για το τρομοκρατικό περιεχόμενο και το πώς το αντιμετωπίζουμε. Οπότε το ζήτημα του ορισμού και πόσο ο ορισμός διαφέρει από χώρα σε χώρα είναι σημαντικό. Ας απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Να διευκρινίσουμε τι είναι παράνομο, τι είναι τρομοκρατικό. Νάταλι Γκρίσπεκ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. που ήρθατε σε αυτή την πρώτη συζήτηση της καινούργια πρόταση κομισιών για την απόσυρση του τρομοκρατικού περιεχομένου online. Ίσως δεν θα καταφέρω να μείνω για να ακούσω και την απάντησή σας, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσεις, ούτε οι σκιώσεις ηγητές δεν καταφέρουν να είναι εδώ. Εν πάση πτώση, εγώ πρόεδρος της Επιτροπής ε, για τον Λόγο της Τρομοκρατίας και ως μέλος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, ε, χαίρομαι για αυτή την πρόταση. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση και θα συνεργαστούμε με την κυρία Στίβενς. Πρόκειται για ένα στρατηγικό νομοθετικό κείμενο μεγάλη σημασίας. βασίζεται σε ένα πολύ ισορροπημένο νομικό καθεστώς και μιλώντας για ισορροπία πρέπει να συνεργαστούμε για να βρούμε ακριβώς αυτή την ισορροπία. Μια ισορροπία που θα είναι δυσεπίτευτη και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να δημιουργηθούν υπόνοιες λογοκρισίας, υφήμωσης. Ίσως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τις μικρές πλατφόρμες να εντοπίσουν αυτό το τρομοκρατικό περιεχόμενο. Έχω μία ερώτηση. Αν θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για τη σύνδεση του θέματος με την Ευρωπόλ. Μέσα στην Ευρωπόλ υπάρχει μια υπηρεσία εντοπισμού τρομοκρατικού περιεχομένου στο ίντερνετ. Ζητώ συγγνώμη αν χρειάζεται να φύγω νωρίτερα. Ευχαριστώ. Okay, thanks, Natalie. Ευχαριστώ, Νάταλη. Ωραία. Σεσίλ Κιέγγε. Oh, ε, Κατερίνα. Κατερίνα. Εσύ πρώτη. Ναι, ναι, Κατερίνα. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν ε, παρούσα, αλλά σήμερα, όπως συχνά συμβαίνει, συνεδριάζουν και η ΛΥΜΠΕ και η ΚΟΝΤ, που έπρεπε να παρέμβω για ένα θέμα που ήταν ε, υπό εξέταση. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Κέγκε που ε, πολύ ευγενικά θέλησε να πάρω πρώτο το λόγο γιατί με τον Επίτροπο έχουμε ήδη συναντηθεί επανειλημμένα για αυτά τα ζητήματα. Έχουμε συζητήσει για το πρόβλημα που συνδέεται με την επικραμική διάδοση προγραμμάτων που παροτρύνουν ε, στη βία. Έχουμε μιλήσει για την αφαίρεση τέτοιων περιεχομένων. Μιλήσαμε για την ανάγκη και θέλω να το να εξασφαλίσουμε κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με την αφαίρεση του περιεχο... περιεχομένου. Αλλά η ερώτηση που εγώ θέλω να υποβάλω στην προσοχή του Επιτρόπου King, τον οποίο ευχαριστώ γιατί πάντοτε είναι παρόν σε αυτό το είδος τα θέματα, τόσο στην Επιτροπή Λίμπε όσο και στην Επιτροπή για την Τρομοκρατία, αφορά μια άλλη πτυχή που είναι πολύ λεπτή. Ε, ε, στις επόμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές ε, έρχονται και ρωτώ πώς σκοπεύει να δουλέψει η Κομισιόν για να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές μέσω των δικτύων για τις εκλογές, για τέτοια σημαντικά θέματα ε, γιατί πώς θα προστατέψουμε λοιπόν την δημοκρατία από αυτού του είδους τις ε, παρεμβολές. Ε, πολύ σημαντικό. το ανέφερε η Διεπίτροπο στην εισήγησή του, αλλά θα επεκταθεί. Σεσίλ, εσύ τώρα. εντάξει, καλύφθηκες. Και στην προηγούμενη συνεδρία ε, τελικά ε, δεν μπόρεσε να υποβάλεις πλήρως την ερώτησή σου. Θέλω να πω ότι είστε μία από τις ευγενέστερες στην Επιτροπή. Ε, Μίχαλ Μπόνι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την σαφή σας παρουσίαση. για την παρουσίαση και για τις προσπάθειες που κάνετε. Με αυτήν την ευαισθησία που αναφέρατε σήμερα για τις μικρές πλατφόρμες, για τους αφείς κανόνες και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλά θέλω να πω κάτι για τις εκλογικές δραστηριότητες στη χώρα μου. Έχουμε στην προοπτική ε, έχουμε μάλλον ε, σε δύο εβδομάδε τοπικέ και περιφερειακές εκλογέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σαφείς κανόνες στο ευρωπαϊκό επίπεδο ε, σε σχέση καταρχάς με τη διαφάνεια και δεύτερον τη λογοδεσία όλων των πολιτικών διαφημίσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όχι μόνο λόγω της Ρωσίας, βεβαίως, αλλά γιατί και από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που θέλουν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεύτερον, χρειάζεται να δώσουμε πολύ ισχυριότερα και συγκεκριμένα εργαλεία για να καταπολεμηθούν οι ψευδείς ειδήσει, που πράγμα που δεν είναι πολύ εύκολο. Αλλά νομίζω πως κάποιο είδους συνεργασία με τις πλατφόρμες, με τις εταιρείες ε, είναι πολύ σημαντική ε, και στην Πολωνία για παράδειγμα συζητάμε για κάποιο είδους κώδικα διοντολογίας για τις εκλογές ε, ανάμεσα στους πολίτες, τις εταιρείες, τις ΜΚΟ. Τελευταία μου παρατήρηση που είναι πολύ σημαντική είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ότι κάποια ρομπότ και αυτοματοποιημένες ε, πληροφορίες που προωθούν τη διάδοση σε τεράστια κλίμακα θα περιοριστούν. από την απέτηση ότι ας πούμε το επίσημο εκλογικό περιεχόμενο θα πρέπει να υπογράφεται από τις πολιτικές επιτροπές των κομμάτων, ώστε δηλαδή να μην υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς αυτά τα ρομπότ. Ε, γιατί αυτού του είδους οι τεχνικές δεν φέρουν υπογραφή. Είναι, δεν είναι εύκολο για να συζητηθεί, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση νομίζω. Έχουμε μια ειδική ομάδα, στη δική μου πολιτική ομάδα συστήση, που παρακολουθεί την κατάσταση μέρα τη μέρα. Τι γίνεται με το ε, στο διαδίκτυο, ποιες, ποια είναι η συμπεριφορά διαφόρων ομάδων και νομίζω ότι μετά τις εκλογές που θα γίνουν στις 21 Οκτωβρίου θα είμαστε έτοιμοι με μια έκθεση προς εσάς γιατί είναι, είναι πολύ σημαντική εμπειρία. Με αυτά τα καινούργια δεδομένα. Ευχαριστώ. Άννα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην προσπάθεια αυτή, η προσπάθεια αυτή βέβαια της τρομοκρατίας είναι πάρα πολύ σημαντική και οι ειδικοί συμφωνούν ότι μεγάλο κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι η αντιμετώπιση της προπαγάνδας από ομάδες όπως το Ισλαμικό κράτος. Βεβαίως καλωσορίζω την ιδέα ότι να μπορεί να αφαιρείται το τρομοκρατικό περιεχόμενο πιο γρήγορα, αλλά όπως έχει η πρόταση αυτή τη στιγμή βλέπω και κάποιου κινδύνους. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς εξαιρέσεις για τα ΜΜΕ και καλύτερες ε, κλίδες ασφαλείας ε, γιατί μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά το περιεχόμενο σε διαφορετικές χώρες. Υψηλά πρόστιμα όπως αναφέρθηκε και γρήγορη χρόνη αντίδραση. Εδώ νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Και υπάρχουν χώρες που έχουν καθορίσει το τρομοκρατικό περιεχόμενο πολύ ευρύτερα από ό,τι εμείς. Ελπίζω λοιπόν να το λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό οι πολιτικές ομάδες και να μην ε, τρέξουν να το περάσουν, γιατί αυτά τα πράγματα έχουν συνέπειες. Σας ευχαριστώ κύριε Κίνγκ. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά και ελπίζω να συνεχίσει η βελτίωση της πρότασης. Ευχαριστώ, Χουάν Φερνάντο. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Παρουσιάζεται εδώ την πρόταση της Κομισιόν για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο και αναφέρεται ρητά οι ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάποιες από αυτές τις ανησυχίες σχετίζονται ακριβώς με το ότι ποικίλει το ποινικό δίκαιο των κρατωμένων σε σχέση με το τι εστί τρομοκρατικό περιεχόμενο. Αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω. Έχουμε μια διάκριση η οποία χάνεται στην κρίζα ζώνη μεταξύ τρομοκρατικού περιεχομένου και λοιπού. άλλα πράγματα κάποιοι το θεωρούν ε, μέρος της ελευθερίας της έκφρασης. Ε, π.χ. εκθιασμός ε, της τρομοκρατίας. Καμιά φορά είναι δύσκολο να το διακρίνουμε από τη μουσική τη ραπ ή από κάποιους blogger που αναπτύσσουν τις σκέψεις τους. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν το έχετε σκεφτεί καθόλου. Γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που εκκρεμούν στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια των κατομμύρων. Π.χ. στην Ισπανία υπάρχει ένας ράπερ. Εδώ, στο Βέλγιο που ζήτησε άσυλο στο Βέλγιο γιατί διώκεται για ένα τραγούδι ας πούμε στο οποίο προσέβαλε το στέμα. Και έτσι κατηγορείται για υποκίνηση βίας κατά του στέματος. Ένα, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Θα λοιπόν να το σκεφτείτε αυτό, γιατί έχει εκφραστεί αυτή η ανησυχία στις συζητήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία η Τερέζα. Σας ευχαριστώ και θα είμαι σύντομη. Ήθελα να πω και δεν είχα την ευκαιρία να το πω τις προάλλες στην Επιτροπή για την Τρομοκρατία, αλλά είναι πολύ σχετικό με αυτό που είπε ο Χουάν Φερνάντο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ορισμό του τι είναι τρομοκρατία, γιατί πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ορισμός του τι είναι τρομοκρατία. Και άρα, εφόσον δεν υπάρχει ε, ορισμός, δεν υπάρχει και ορισμός ε, για την παρότρινση, την, ε, τον εκθιασμό στην τρομοκρατία. Ε, στην Ισπανία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί υπάρχει κενό και στην κοινή μας ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσα στο πλαίσιο της ε, ε, προστασίας και των θυμάτων εφόσον υπάρχει έλλειψη της εντολής για την σύλληψη των, των των δραστών, ε, η ταπείνωση των θυμάτων είναι και αυτό ε, ε, αδίκημα. Έχουμε στο Βέλγιο έναν τρομοκράτη στην Γάνδη που με εγκλήματα, που πορεύει σε εγκλήματα αίματος και τώρα μόλις αποκαλύφθηκε πως ακόμα έχει διαπράξει δύο, δύο ακόμα εγκλήματα αίματος και δεν τον επιστρέφουν στην Ισπανία, δεν τον απελάσουν. Ε, ε, είναι λέει ένας πολίτης δεν μπορεί να πάψει να είναι δολοφόνος. Είναι δολοφόνος ακόμα και αν δεν θεωρείται ότι είναι τρομοκράτης πρέπει να επιστραφεί και να δικαστεί. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αυτό υπάρχει λοιπόν και ότι θα πρέπει να το κατανοήσουμε, μάλλον το κατανοούμε καλύτερα μόνο όταν ε, ε, ξέρουμε και ποια είναι τα θύματα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αλληλεγγύη με αυτό και είναι πραγματικότητα ότι δεν μπορούμε να δίνουμε ε, συγχώρες ούτε να γίνεται έτσι τόσο κάτι το κοινό η τρομοκρατία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, επειδή αυτή είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, να σας ρωτήσω τι αντιδράσεις είχατε για την πρόταση αυτή. Αφενός για τους ειδικού ε, που προσπαθούν να κατεβάσουν ε, διάφορες σελίδες. Ε, ξέρουμε ότι η Europol το κάνει ήδη όσοι το ξέρουν αυτό το θέμα και ασχολούνται με αυτό. Και ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Δεν θα εκπλαγούν από τα όσα περιέχει η πρώτη Ο κόσμος δεν, που δεν τα ξέρει αυτά θα κάνει ερωτήσεις όπως αυτές που ακούσαμε για τους ορισμούς και τα λοιπά. Παραδείγματος χάρη παρατηρώ εδώ στη σελίδα 15 μιλάτε για την ε, έκφραση ζωσπαστικών επίμαχων απόψεων κτλ αν δούμε τρομοκρατικό περιεχόμενο μη ισλαμικό, ας πούμε της άκρας δεξιάς, ε, οι υπηρεσίες ε, ασφαλείας ε, γνωρίζω στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Γεροπολ λένε ότι αυξάνεται η παρακίνηση στη βία. Όμως φανίζονται όλο και περισσότερα τέτοια στα κοινωνικά μέσα. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξής. Όταν ε, κάνετε αυτή την πρόταση υπάρχει κάποια ενημέρωση για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε και πόσο πολλά έχετε να κάνετε γιατί ε, βεβαίως ε, εδώ πέρα έχετε κάτι το διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνει η Europol που βεβαίως παρεμβαίνει αμέσως, ε, το οποίο εμένα με βρίσκει σύμφωνο, αλλά βεβαίω όταν βλέπω μια τέτοια πρόταση ε, πρέπει να το πετύχουμε, να πετύχουμε την ισορροπία, να μην απαγορεύουμε πράγματα και να μπλέξουμε. Για πώς ακριβώς ε, λοιπόν θα εξηγήσουμε τις διαχωριστικές γραμμές Συγγνώμη αν το κάνω πολύ φιλοσοφικό, αλλά αν διαβάσει κανεί το περιεχόμενο τη πρόταση είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή η οποία πρέπει να γίνει. Ε, την οποία καλωσορίζω, λέει ο Πίτροπο. Δεν θέλω οπωσδήποτε να βιαστούμε και να μην ε, το εξετάσουμε προσεκτικά ακριβώς για να εξηγήσουμε το τι είναι και τι δεν είναι αυτή η πρόταση. Και έχει σημασία το τι δεν είναι. Δεν ε, προτείνουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να περιγραφεί ως λογοκρισία. Στοχεύουμε ένα συγκεκριμένο είδος περιεχομένου, αλλά θέλουμε να καθοριστεί σαφώς σε ολόκληρη την Ευρώπη με έναν ξαφή ορισμό του τι είναι παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο. Και μετά, αυτό λοιπόν για την κυρία Σίπελ, και μετά να καθορίζουμε τους κανόνες και τις ε, διαδικασίες ε, για να ταυτοποιείται και να κατεβαίνει αυτό το περιεχόμενο. Και οι αντιδράσεις που είχαμε μέχρι στιγμής από ολόκληρη την Ευρώπη είναι θετικές. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ε, αλλά πρέπει ο διάλογος να πάει πέρα από το τεχνικό επίπεδο. Και τα έχουμε εξηγήσει αυτά δημοσίως όσον αφορά τον ορισμό στον οποίο θα επανέλθω. Οι αντιδράσεις που είχαμε από τις πλατφόρμες είναι κυρίως θετικές. Δεν είχαμε κάποια πλατφόρμα η οποία είπε «Α, όχι, αυτό δεν το θέμα». Όπως σας είπα, οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν τους πόρους και βεβαίως θέλουν να προστατεύσουν και την φήμη τους. Αυτό το οποίο μας ζήτησαν είναι να είμαστε πιο ξεκάθαροι όσον αφορά τι κανόνες. Από τη ΣΥΠΑ είχαμε αρνητική αντίδραση. Μας εξήγασαν και πάλι χτες όταν είχε πάει ο Δημήτρης Αδάμουπλος ότι δεν τους αρέσει. Θεωρούν ότι στοχεύει τις εταιρείε τους. Εμείς τους εξηγήσαμε ότι δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Απλά για μια συγκεκριμένη κατηγορία περιεχομένου. Λένε ότι είναι κατά της ε, πρώτης ε, τροπολογίες του συντάγματος. Ε, εμείς λέμε ότι δεν είναι ζήτημα ελευθερίας λόγου αλλά να υπάρχει η πιθανότητα, όπως είπε η κυρία Σίπελ, να αστυνομεύεται το παράνομο περιεχόμενο. Εάν ήταν παράνομο σε ένα φυλάδιο στο δρόμο, γιατί δεν είναι παράνομο επειδή είναι στο διαδίκτυο. Εμεί δεν θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι εκτός αστυνόμευσης ε, το διαδίκτυο. Πρέπει λοιπόν να το πούμε αυτό λένε ότι μπορεί να πλήξει την καινοτομία με κάποιον τρόπο, αλλά δεν μπορούν να μας εξηγήσουν το γιατί. Να προσπαθεί να ε, δει το θέμα του διαδικτύου. Εγώ δεν βλέπω να εμποδίζεται καμία καινοτομία πριν από την καινοτομία της ε, τρομοκρατίας. Οπότε έχετε δίκιο ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε τα πράγματα στο κοινό και πιθανώς διεθνώς. Αλλά αυτά δεν με αποθαρρύνουν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα και ελπίζω μαζί σας να μπορέσουμε να βελτιώσουμε. Τα ζητήματα αυτά. Βεβαίω ε, σημαίνει ότι θα χρειαστεί χρόνος ε, και προσπάθεια και αισθάνομαι κάποια ενοχή που συζητάω να ασχοληθείτε και με αυτό, αλλά είναι τόσο σημαντικό και τόσο επίγον που νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Είδαμε το ζήτημα των ορισμών ρητός και μπορείτε να μας βοηθήσετε να μας ρωτήσετε για να δούμε αν τα έχουμε πετύχει, αν τα έχουμε κάνει σωστά. Ε, ξεκαθαρίζουμε ερτός πως το περιεχόμενο το οποίο διαδίδεται για εκπαίδευση, για έρευνα από δημοσιογράφους κτλ. Εξαιρείται. Αν θέτε να το κάνουμε πιο σφιχτό, αλλά προσπαθούμε να είμαστε σαφείς. Μετά καθορίζουμε το τρομοκρατικό περιεχόμενο ακριβώς προσπαθώντας να βρούμε τον ορισμό που έχουν ε, διάφορες ε, πλατφόρμες. Έχουμε γράψει λοιπόν εμείς έναν ορισμό που θα γίνει ο ορισμός στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εάν συμφωνήσετε. Και βασίζεται στην οδηγία καταπολέμησης τρομοκρατίας ε, και σε κάποια ομάδα που έχει καθορίσει ο ΟΗΕ. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς για το τι εννοούμε και το τι δεν εννοούμε στο περιεχόμενο. Ακριβώς για να υπάρχει και μια σύνδεση με κάποιους οργανισμούς, με κάποιες οργανώσεις που γνωρίζουμε διεθνώς ότι ε, παράγουν τέτοιο περιεχόμενο. Και εδώ πέρα αυτό είναι μια πρόκληση, γιατί έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο ο τζιχαντισμός που μας απασχολεί, υπάρχουν και άλλες μορφές ε, που δεν τις καθορίζει πάντα ο ΙΕ. Αυτή είναι λοιπόν η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και αν τα καταφέρουμε νομίζω ότι θα ανταποκριθούμε σε πολλές από τις ανησυχίες που ακούστηκαν γιατί εξηγεί το γιατί προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να υπάρχει ένας διασυνοριακός ορισμός και έτσι μπορούν τα κράτη-μέλη να καταλήξουν σε κάποιες αποφάσεις και να μην ε, επομίζονται πλέον το βάρος μικρές και μεσαίες πλατφόρμες ε, στις οποίες αυτή τη στιγμή ρίχνουμε το βάρος μέσω των όρων χρήσης. Ε, εγώ θεωρώ λοιπόν ότι έτσι τους βοηθούμε. λοιπόν και εάν το πετύχουμε αυτό νομίζω ότι έτσι θα εξηγήσουμε το γιατί αναλάβουμε δράση εδώ και όχι σε κάποιον άλλο τομέα. Μερικές φορές έχουμε αιτήματα να δούμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα της ρητορικής μίσους. Α, δεν είναι αυτή η πρόταση αυτή. δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα με πανευρωπαϊκή νομοθεσία. Γιατί υπάρχουν ιστορικές διαφορές, νομικές διαφορές που είναι δύσκολο να συμβιβαστούν. Αλλά θεωρώ ότι γνωρίζουμε το τι είναι τρομοκρατικό περιεχόμενο και υπάρχει συνένεση στην Ευρώπη, στις διάφορες χώρες που θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε έναν ε, ορισμό. Για το θέμα των ε, μέσων ε, που θα απαιτηθούν από τα κράτη-μέλη, στόχος είναι να υπάρχει μια εθνική ομάδα παραπομπής ίντερνετ σε κάθε χώρα. Προτείνουμε κάτι τέτοιο για να υπάρχει δυνατότητα να αυτοποιηθούν αυτά και επίση θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσφυγή και δικαστικής προσφυγή και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αν είναι δυνατόν ο ρόλος της ε, Europol που κάνει πολλή δουλειά για να βοηθήσει διάφορες πλατφόρμες που έχουν ε, μεγάλο απόθεμα υλικού Οπότε περιλαμβάνουμε ακριβώ ότι μπορεί να γίνει στο επίπεδο των διεκτικών αρχών, να καλύψουμε την συνεργασία με την Europol, ε, η οποία θέλουμε να εμπλέκεται, αλλά το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, η Europol δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Δεν μπορεί δηλαδή να επειδή της τις ε, δικαστικές ε, είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι περιορισμός, ε, μπορεί να συντονίζει τις εθνικές αρχές. Όσον αφορά ακριβώ το θέμα της ασφάλειας των εκλογών, είπα πριν φτάσετε το τι προσπαθούμε να κάνουμε σε γενικές γραμμές, δηλαδή να δούμε τις παραδοσιακές κυβερνοεπιθέσεις σε φυσικές υποδομές κτλ. και εκεί πέρα ακριβώ πρέπει να ε, ενισχύσουμε την καλή δουλειά που κάνουν οι ειδικοί της ε, κυβερνοεπιστήμης και να αυξηθούν και οι κανόνες ε, προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως είπε και η κυρία Γιώργα και να αλλάξουν οι κανόνες χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών κομμάτων για να υπάρχει δυνατότητα κυρώσεων εάν δεν προστατεύουν τα δεδομένα που έχουν αλλά Υπάρχουν διάφορα ενδιάμεσα ζητήματα που είναι τα δυσκολότερα. Ε, σχετίζονται ακριβώς ε, με τέτοια ζητήματα χειραγωγήσεις. Και εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Επίτροπο Γκαμπριέλ ε, φτιάξαμε έναν πρώτο διεθνή κώδικα συμπεριφορά. Συνεργάζονται οι πλατφόρμες μαζί μας για να δούμε κάποια ζητήματα που μας ανησυχούν. Ε, διαφημίσεις, ε, περιεχόμενο προωθημένο, τα bot, ε, διαφάνεια για εξωτερικούς ερευνητές, για να δουν ιστορικά υπερβάθες του παρελθόντος κτλ. Και έτσι είπαμε ότι εντάξει, καλά το κάνουμε στιγμή, αλλά πρέπει τώρα να καθορίσουμε κάποια μετρήσιμα παραδοτέα, κάποιους στόχους, για να μπορέσουμε ακριβώς να μετρήσουμε την πρόοδο μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί η συνεργασία. Από την άλλη πλευρά, έχουμε πει ότι για τα πολιτικά κόμματα, το έχουμε βάλει αυτό στις συστάσεις, θα θέλουμε τα κράτη-μέλη να είναι σε επαφή με τα πολιτικά κόμματα, να ενθαρρύνουν τα πολιτικά κόμματα τα ίδια να λάβουν κάποια βήματα διαφάνειας για το τι ξοδεύουν στο διαδίκτυο για τις διαφημίσεις. Νομίζω λοιπόν πως έτσι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο για ένα ζήτημα το οποίο αναγνωρίζω είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Σας ευχαριστούμε. Ε, το που λέμε εμείς είναι αν θέλεις να γίνει κάτι ρώτα κάποιον ο οποίος είναι απασχολημένος. Η πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ περίπλοκη και μια ολόκληρη πρόκληση. Είναι μια, ένα τεράστιο βήμα, ένα, μια νομοθετική πράξη που χρειάζεται πολλή ενημέρωση, του κοινού είναι μια αλλαγή συστήματος μοντέλου. Εμείς θα βιαστούμε. Μπορώ να πω κάτι ακόμα γι' αυτό. Συμφωνώ για όλα αυτά, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να το παρουσιάσετε έτσι. Μήπως και κάποιος πιστεύει ότι προσπαθούν να φάμε μια μπουκιά πιο μεγάλη από αυτή που μπορούμε να μασίσουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι στα μέτρα μας. Θα ξεκινήσουμε τον ορισμό και αν πετύχουμε στον ορισμό όλα τα άλλα θα πέσουν σαν όριμο φρούτο. Συμφωνώ. Απλά έχουμε τρεις μήνες μόνο. Τέλος πάντων, τα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είστε η πιο ικανή επιτροπή, λέει ο Επίτροπος. Έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και οι και οι Αν δείτε πόσα θέματα δουλεύουμε παράλληλα, κάνουμε γρήγορους διορισμούς, οι άνθρωποι ξεκινάνε να δουλεύουν αμέσως. Την περασμένη εβδομάδα μόλις διορίσαμε ένα μεγάλο αριθμό εισηγητών για διάφορα θέματα που εκκρεμούν. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μέρα ήταν πολύ έντονη, δύσκολη. Χαίρομαι που σας είχαμε κύριε Επιτρόπο μαζί μας. Ευχαριστούμε Χέλγα που έδωσε το αναρκτήριο Θα τα ξαναπούμε για αυτό το ζήτημα. Συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και σας κύριε Επίτροπε. Uh, Συνάδελφοι, ξεκινάμε το σημείο 14. Καλωσορίζω θερμά τον ειδικό απεσταλμένο της ε, είπα της αρμοστίας του ΕΕ για τους πρόσφυγες για την κατάσταση στην Κεντρική Μεσόγειο, Vince Κοσετέλ και τον Ευγένιο Αμπρόζη, Περιφερειακό Διευθυντή του Περιφερειακού Τμήματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας συγχαίρω για την πολύ ε, καλή δουλειά που κάνετε. Έχουμε έρθει σε επαφή για πολλά από αυτά τα θέματα ε, και φέτος το καλοκαίρι τελευταία με τον κύριο Κοσετέλ και τον κύριο Αμπρόζη. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά που, εξαιρετική δουλειά που κάνει. Μιλήσαμε και με τον ίδιο κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Έχουμε πάρα πολλά θέματα για το άσυλο, για τις επιστροφές, για την υπηρεσία, την ΕΑΣΟ κλπ. Η συνάντηση αυτή μεταδίδεται και μέσω του ίντερνετ. Ε, οπότε μην ανησυχείτε, δεν βλέπετε πολλούς εδώ μπροστά σας, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που μας βλέπει από το ίντερνετ. Συμπέρασμα του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ε, προτάσεις για το άσυλο από την Κομισιόν, Έχουμε πολλά καινούργια στοιχεία και οι δυο σας έτσι κι αλλιώς βλέπετε πολύ κοντά την κατάσταση στη Μεσόγειο. Όλοι μας, ε, όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, γνωρίζουμε τον κεντρικό ρόλο που παίζεται. Το, το απόγευμα ήδη συζητήσαμε για πολλές ώρες αυτά τα θέματα. Έχουμε ήδη καθυστερήσει Οπότε δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα ζητήσω καταρχήν, θα καταρχήν από το Βενσό να πάρει το λόγο για μία εισαγωγή. Και ο Εουτζένιο θα πάρει το λόγο μετά. Ευχαριστώ την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την πρόσκλησή σας να έρθω εδώ και για την πολύ καλή συνεργασία με τον ΟΗΕ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί στη, κάποιοι από εσά στείλατε μια επιστολή για το τι, που ρωτούσατε τι ακριβώς κάνουμε στη Λιβύη ή τι δεν κάνουμε στη Λιβύη. Θα σας στείλουμε μια απάντηση επίσημα, θα μιλήσω και εγώ για το θέμα. Καταρχήν να σας επενέσω για την πολύ καλή δουλειά που κάνατε στις διαπραγματεύσεις για την μεταρρύθμιση του ασύλου, υπογραμμίζοντας ότι για μας η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου είναι ύψης της προτεραιότητας. Δουλεύουμε για αυτό το πακέτο από την αρχή με ε, εξειδικευμένη γνώση βοηθήσαμε το Συμβούλιο να αναπτυχθεί ο μηχανισμός περιφερειακής, ε, περιφερειακών ε, αποβιβάσεων, ε, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου χρειάζεται ασφαλώς ε, μεταρρύθμιση, αλλά οι πλατφόρμες δεν είναι υποκατάστατο. Δεν είναι έτσι κι αλλιώς ε, δυνατό να ζητούμε από τους εταίρους μας να κάνουν πράγματα για τα οποία εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Οπότε υπήρξαν παρεξηγήσεις ε, και εδώ και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πολλές ήταν οι φωνές που υψώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να μοιραστούμε την ευθύνη στις δύο πλευρές τη Μεσογείου. Δεν, στόχος δεν είναι να μεταφερθεί η ευθύνη από τη μία όχθη τη Μεσογείου στην άλλη. Λιβύη, δεν έχουμε πολύ πρόοδο. Από το τελευταίο φορά που συναντήκαμε ξέσπασε ακόμα ένα γύρος ε, σύραξης. η Η Τρίπολη, οι, ε, οι οργανώσεις της ε, Τρίπολης δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Η κατάσταση παραμένει στα σημεία. κάποια κέντρα κράτησης έχουν κλείσει, κάποια άλλα ανοίγουν. Ε, μετανά, οι ετούντες άσυλο πολλές φορές ξεφεύγουν, αποδρούν ε, άλλοι χάνονται τελείως, η πρόσβαση είναι περιπλοκή. Μπορώ να σας πω ότι κάθε φορά που η ακτοφυλακή ε, πιάνει ε, άτομα που προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη και τα επαναφέρει στις πλατφόρμες στην Λιβύη, χάνουμε τα ίχνη τους δεν είμαστε παρόντες. Καμιά φορά στέλνουμε κάποιον από τους εταίρους μας, αλλά όχι συστηματικά. Το πρόβλημα έτσι κι αλλιώς δεν είναι με τις αποβιβάσεις, γιατί εκεί μένουν δύο-τρεις ώρες. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται μετά, σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους. Πρέπει να δούμε τι γίνεται τις επόμενες 24-48 ώρες μετά την αποβίβασή τους. Το σύστημα τη αποβέρσης στη Λιβύη δεν μπορεί να κρυθεί με βάση τις πρώτε δύο ώρες. Κανονικά αυτά τα άτομα μεταφέρονται σε κέντρα κράτηση, ε, μερικοί όμως χάνονται στο δρόμο. Ε, δεν είναι ότι ξεφεύγουν, απλά πολλούνται σε δουλεμπόρους, σε εκμεταλλευτές κλπ. Πολλοί λοιπόν χάνονται κατά τη μεταφορά τους στα κέντρα κράτησης. Εκεί υπάρχουν επίσημα τρία κέντρα κράτησης. Στη Λιβύη, συγγνώμη, ε, πέντε στην Τρίπολη, δέκα στη Δύση, πέντε στο Νότο, ε, δεν είναι τρία, είναι περίπου τριάντα. Ε, έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε τρία κέντρα τη βδομάδα, στην Τρίπολη, στη Δύση. Δεν μπορούμε να καλύψουμε λοιπόν όλα τα κέντρα και να είμαστε πάντου παρόντες. Προφανώς η διάσπορα, ε, η, διασπο, η, η, οι Λιβανέζοι που ζουν στην Ευρώπη διαμαρτύρονται, έχουν χάσει επαφή με πολλούς συγγενείς τους. Εμείς όμως δεν έχουμε πρόσβαση πολύ συχνά και ακόμα και όταν έχουμε πρόσβαση δεν βρίσκουμε πάντοτε τους ανθρώπους που περιμένουμε εκεί, έχουν ήδη μετακινηθεί και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και θέματα ασφάλειας του προσωπικού μας με πολλά από τα κέντρα κράτησης. Είχαμε συζητήσει την δυνατότητα μια, ενός ενδιάμεσου κέντρου ε, Υπάρχει ένα τέτοιο κέντρο χιλίων ατόμων, ε, δεν έχει ανοίξει όμως, υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα. Αυτό είναι ένα κέντρο μεταγωγής. Ε, δυστυχώς δεν έχει ανοίξει, η κατάσταση παραμένει στάσιμη. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση για τις ε, Για τις επαφές με τις ε, χώρες της Βορειάς Αφρικής να σας πω ότι ε, θα πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στους μηχανισμούς που υπάρχουν σε κάθε μία από αυτές τις χώρες. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα συνολικό σχέδιο. Το Μαρόκο, την Ισία, Αλγερία και Αίγυπτος. Ε, εκεί εργαζόμαστε σε αυτές τις χώρες από το 50 έχουμε γραφεία. Υπάρχουν δυνατότητες αποβίβασης ατόμων ε, που εντοπίζονται στη θάλασσα με διαφορετικά συστήματα σε κάθε χώρα. Τα συστήματα αυτά δεν είναι τέλεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργούν. Υπάρχουν κάποιοι υποτυπώδεις μηχανισμοί υποδοχής και θα πρέπει πάνω σε αυτούς να οικοδομήσουμε έτσι ώστε τελικά να διέπονται από το κατάλληλο διοικητικό και νομικό πλαίσιο. Πράγμα που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται πολιτική βούληση για να γίνει αυτό. Έχουν υπογράψει τη σύμβαση του 1951, αλλά χρειάζεται χρόνος ε, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε υπεύθυνα με αυτές τις χώρες. Δεν είναι δυνατόν να, αλλάξουμε από τη μια μέρα, να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε να γίνουν πολύ ε, μεγαλειώδεις ε, και πανηγυρικές δηλώσεις. Τέλος, ακούω πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες που λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλά πράγματα στο Μαρόκο, στην Τινησία, στην Αίγυπτο, γιατί δεν κάνετε αυτό ή δεν κάνετε εκείνο. Το επίπεδο χρηματοδότηση στην Αίγυπτο είναι 42%, στο Μαρόκο 23%, στην Τινησία 16%. Οπότε ήδη δεν έχουμε αρκετή αλληλεγγύη μέσα στην Ευρώπη, πολύ λιγότερο μάλιστα με τις χώρες εκτός Ευρώπης. Σε όλες αυτές τις χώρες περικόπτουμε τα προγράμματά μας μόνο το 15% των προσφύγων δέχονται βοήθεια στο Μαρόκο, 20% των προσφύγων στην Αίγυπτο, σε σχέση με το 40% που ήταν πέρσι. Οπότε η συνδρομή μας μειώνεται. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όλο και πιο ευάλωτοι, όλο και πιο πιθανό να μετακινηθούν σε μια γειτονική χώρα. Οπότε μην εκπλαγούμε. Δεν μιλούμε για συγκράτηση, <laughs> αλλά αν θέλουμε να τους δώσουμε μια εναλλακτική λύση έναντι της μετανάστευσης, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες σοβαρά. Με προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή η συνδρομή που παρέχουμε είναι πολύ χαμηλότερη από το επιθυμητό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που μας στηρίζετε. I do want to say to you, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε να σας ξαναδούμε λόγω αυτών των πολύ σημαντικών θεμάτων που μας αναφέρετε, αλλά χρειάστηκε στη σημερινή μέρα να σας τριμώξουμε στο τέλος. Ελπίζω να μην σας πειράζει να ξαναέρθετε. Δεν θέλω να χάσω τους τρεις βουλευτές που είναι εδώ. Οπότε, Τζένι, αν μπορείς να είσαι πιο σύντομος για να προλάβουμε να ακούσουμε και ερωτήσεις. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαστε ευτυχείς που είμαστε σήμερα εδώ και να συνεχίζουμε το διάλογο μαζί σας για το θέμα της Κεντρικής Μεσογείου και τον μηχανισμό αποβιβάσεως που περίγραψε ο Βενσό. Βεβαίως, ε, και σύμφωνα με όσα είπε μόλις ο Μεσά. απλά να προσθέσω ένα-δυο ε, προβληματισμούς. Καταρχάς, το δικαίωμα στην αποβίβαση ε, είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να επαναλάβουμε το παράδοξο της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη όσον αφορά την κεντρική Μεσόγειο και το θέμα των αφήξεων και της αποβίβασης. Το παράδοξο είναι ότι ο αριθμός των αφήξεων έχει μειωθεί πολύ σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και το προπροηγούμενο πάντοτε ισχυριζόμασταν ότι οι αφήξει ε, ακόμα και στην αιχμή του το 2015 η αφήξει ήταν εύκολο να τις διαχειριστούμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Δηλαδή εφόσον μπορούσαμε να τι διαχειριστούμε όταν έφταξε ένα εκατομμύριο κόσμο, ε, τόσο πιο εύκολο είναι και να χειριστούμε τις 80.000 κόσμο που έχουν φτάσει στην Ευρώπη, δηλαδή σε 40% λιγότερο από πέρσι. Όμως έχουμε διπλό, διπλάσιο αριθμό θανάτων στην Μεσόγειο. Δηλαδή είναι πιο επικίνδυνο τώρα το να διασχίσει κανείς τη Μεσόγειο από ό,τι πριν. Και έχουμε και αντιδράσεις στην Ευρώπη που είναι πολύ πιο έτσι, και αποσπασματική από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Ε, τεράστια αύξηση στο ποσοστό θανάτων λοιπόν. Πολλά μέτρα έχουν ληφθεί για να καταστεί δυσκολότερη η έρευνα και η διάσωση στη θάλασσα λόγω της πάυσης της δράσης το σκάφος του ΣΜΚΙΟ που μέχρι πρόσφατα και μέχρι ότου που μπορούσαν να λειτουργήσουν ήταν υπεύθυνη για την διάσωση περίπου του 40% των όσων σώζονται στην Μεσόγειο. Λήφθη απόφαση ότι είναι εγκληματική εργασία κάποιων που έχουν σώσει ζωές. Και πρέπει να σας πω ότι με μεγάλη ανησυχία βλέπουμε το γεγονός ότι σε κάποια χώρα της Ένωσης ακόμα και η ανθρωπιστική βοήθεια προς έναν άνθρωπο, έναν μετανάστη που έρχεται ε, πλέον θεωρείται αδίκημα. Και άρα το σύστημα είναι πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν θα επιμείνω για τα όσα ήδη αναφέρθηκαν για τον μηχανισμό αποβίβασης που αναφέρθηκε. Απλά να πω ότι η ιδέα είναι να μην αντικατασταθεί με κανένα τρόπο αυτό που θα πρέπει να συμβεί μέσω της έγκρισης και της εφαρμογής του κοινού συστήματος ασύλου. Ο μηχανισμός που συζητάμε είναι ένας μηχανισμός για να καλυφθεί το κενό μιας άμεσης ανησυχίας και προβλήματος που έχουμε, δηλαδή ένας σωστός μηχανισμός για αποβιβάσεις, αλλά και για ε, την ε, διεκπαιρέωση των τυπικών διαδικασιών των όσων σώζονται και βοηθούνται. Αυτό όμως μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν τα κράτη-μέλη ε, μοιραστούν τις ευθύνες καταλήλως μεταξύ τους, ώστε μετά ο διάλογος με τη Βόρεια Αφρική και τη δική του συμβολή ώστε να βρεθεί μια λύση στη Μεσόγειο να μπορεί να υπάρξει. Εφόσον δεν υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη, τότε και καμία βορειοαφρικανική χώρα δεν θα προβεί σε συζήτηση για οποιοδήποτε περιφερειακό μηχανισμό. Θα συνεχίσουν όπως μέχρι τώρα, όπως είπε και ο Βενσό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι ενώ ζητάμε από άλλε χώρε στην Βόρεια Αφρική να μα βοηθήσουν εμά στην Ευρώπη σε αυτήν την κατάσταση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι κάνουν ήδη. Ήδη κάνουν έρευνα και διάσωση και αποβίβαση και βοηθεία προς αυτού που ε, σώζονται. Σε λίγα λεπτά η διερμηνία θα σταματήσει. Γι' αυτό θα ήθελα η κυρία Κέγκε να μπορέσει να υποβάλει την ερώτησή της. Υπάρχουν πολλοί αγγλόφωνοι εδώ, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι αγγλόφωνοι. Εντάξει, θα προσθέσω μετά. Να ακούσουμε λοιπόν την κυρία Κέγκε γιατί θα φύγουν οι διερμηνείς μας. Σεσίλ, θέλεις να θέσει την ερώτησή σου τώρα. Και μετά η κυρία Σπινέλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Κλοντ. Είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή και κυρίως καθώς η Ιταλία, η χώρα μου, κάνει κάτι πολύ θεαματικές δράσεις εντό εισαγωγικών που θέτουν υπό ασφισβήτηση τις αρχές τις οποίες εμείς στηρίζαμε μέχρι τώρα, δηλαδή τη διάσωση των ανθρώπινων ζωών δύο ερωτήματα. Πρώτο, ε, ξέρω ότι προωθείτε ένα project περιφερειακών πλατφορμών και έτσι τα κράτη ε, δεν χρειάζεται, δεν φέρουν πια την ευθύνη, μετακινούνται τα σύνορα προς τα νότια της Ευρώπης. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να επανέλθουμε στην εργασία πάνω στην ευθύνη και στην μοιρασιά της ευθύνης και την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Τελευταία μου ερώτηση για τις ΜΚΟ. Και εγώ είμαι σε τέτοια ιδέα γιατί 11 ΜΚΟ ήταν υποψήφιες για ο βραβείο Ζαχάροβ εδώ στο Κοινοβούλιο. Θεωρώ πως πρέπει να ενισχυθεί η δράση έρευνας και διάσωσης. Χρειαζόμαστε ακριβώς αυτές τις ΜΚΟ που πρέπει να επιστρέψουν για να συνεχίσουν το έργο τους. Σας ρωτώ, Ποιε είναι οι δικές σας προβλέψεις μακροπρόθεσμες προτάσεις, γιατί μέχρι στιγμής μιλάμε μόνο για μια βράχη χρόνια προσέγγιση μακροπρόθεσμα, Ποιε είναι οι προτάσεις σας. Ευχαριστώ. Σεσίλη Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ και τους ε, δύο μιλητές, ε, τον κύριο Κοσετέλ και τον κύριο Αμπρόζη, για τη σημαντική τους συμβολή στη σημερινή συζήτηση. Ζητώ συγγνώμη γιατί μάλλον θα πρέπει να φύγω πριν να ακούσω τις απαντήσεις σας, αλλά θα τις ακούσω στο διαδίκτυο. Εσείς κύριε Κοστέλη είπατε κάτι που, που, με εντυπωσίασε πολύ πριν από κάποιο καιρό. Πώς θα εξηγήσουμε στην επόμενη γενιά ότι αφήσαμε όλους αυτούς τους μετανάστες να πεθάνουν γιατί δεν βρήκαμε συμφωνία για το πώς θα επεξεργαστούμε τα αιτήματα ασύλου του και το πώς θα μοιραστούμε τις ευθύνες. Και εγώ κάθε μέρα να ρωτιέμαι πώς θα το εξηγήσουμε στις επόμενες γενιές. Πώς θα εξηγήσουμε και την προσπάθεια ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τα βάζει όλα στο, στις αναχωρήσεις, την εξωτερήκευση του ασύλου και κυρίως σε σχέση με τις πλατφόρμες στις χώρες που είπατε. Όχι τη Λιβύη, αλλά άλλες χώρες. όπου θα μπορούσε ίσως να λειτουργήσει ένα μηχανισμός. Αυτό που εγώ αναρωτιέμαι είναι, υπάρχει το αρνητικό, υπάρχει το αρνητικό μοντέλο του Νίγηρα που το καιρό του μας παρουσιάστηκε ως μέγα project ε, που θα έλυνε τα προβλήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να επανεγκαταστήσει έναν επαρκή αριθμό μεταναστών. Δηλαδή, μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να δημιουργηθούν κέντρα εκτός Ευρώπης χωρίς να υπάρχουν εγγύησεις, αλλά πραγματικές εγγύησεις, όχι λόγια για επανεγκατάσταση. Εντάξει, έχω και άλλες πολλές ερωτήσεις, αλλά και εγώ είμαι πολύ απελπισμένη. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα. Ο Χαν Φερνάντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Βινσάν Κοζελέ και ο Τζένι Αμπρόζη που είστε εδώ. μεγάλη μέρα σήμερα, δεν έχει τελειώσει η συνεδρίασή μας. Αύριο στις 9 ξαναρχίζουμε. Αλλά πιστέψτε με, οι λίγοι που είμαστε εδώ και που έχουμε επιβιώσει, ε, είμαστε ήδη προσελητισμένοι, δεν χρειάζεται να μας προσελητήσετε. Το πολιτικό θέμα είναι ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα, τεράστια απόσταση ανάμεσα στα στοιχεία και στην αντίληψη που υπάρχει. Πριν από λίγο ακούσαμε τον κύριο Βραμόπουλο στο διευθυνμένο διάλογο. Ναι, ευχαριστούμε για το διευθυνμένο διάλογο, αλλά από εδώ ακούσαμε ερωτήσεις που ε, ε, κατέδειξαν ε, σαφώς πόσο τεράστιο είναι το, το, η, απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και την αντίληψη του τι ισχύει. Σήμερα το πρωί κάναμε συζήτηση για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Και υπευλήθη ερώτηση προς τον Επίτροπο Αβραμόπουλο. Δεν είναι αλήθεια ότι αν ανοίξουμε το παράθυρο για, τα, για νόμιμους μετανάστες, αυτό θα ενθαρρύνει και τους την παράνομη μετανάστευση, την λαθρομετανάστευση. Πραγματικά αυτή είναι μια πολύ ευρέως δεδομένη άποψη που την εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί. Χρειάζεται μεγάλη, πολλή ενέργεια ανάμεσα σε, και συνεργασία ανάμεσα σε εσά και εμάς εδώ που, που ήδη, ε, όπως σας είπα, έχουμε προσελετιστεί. Επίσης ακούσαμε μια ερώτηση προς τον Επίτροπο Αβραμόπουλο που παρέμεινε αναπάντητη. Πόσοι από αυτούς τους λαθρομετανάστες που έρχονται στην Ευρώπη επιστρέφονται στα αλήθεια, γιατί η αντίληψη που επικρατεί είναι ότι έρχονται εκατομμύρια και κανένας δεν επιστρέφεται. Για πείτε μας νούμερα. Νούμερα. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε να διαβάσουμε το μήνυμα ότι η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική, ότι δεν είναι αλήθεια ότι ο αριθμός αυτών που έρχονται λαθρέα είναι τόσο τεράστιος, ενώ αυτοί που επιστρέφονται είναι ελάχιστοι. Εάν μας βοηθήσετε λοιπόν σε αυτό να καταπολεμήσουμε, να καλύψουμε αυτές τις, αυτή την απόσταση, θα έχουμε καταφέρει κάτι για να αλλάξει η κατάσταση αυτή, η οποία είναι πραγματικά παράδεκτη. Ευχαριστώ.